colleagues. Welcome. Συνάδελφοι, καλώς ορίσατε. Παρακαλώ καθίστε όλοι. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Καταρχάς έχουμε τις, ε, τα σχέδια αποφάσεων της συνεδρίασης των συντονιστών της 31ης Σεπτεμβρίου. Είναι, ε, ε, συγγνώμη, της 30 ε, Σεπτεμβρίου υπάρχουν όλα ε, στα, ε, στους φακέλους σας. Η συναδρίαση είναι, διαδίδεται στο διαδίκτυο και είναι και άνευ χαρτιού. Έχουμε την Επιτροπή Έρευνας άρθρο 4,1. Ονόματα και ατόμα δεν μπορούν να δημοσιεύονται. Γι' αυτό και... Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 15 Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο και της 30 Σεπτεμβρίου θα διορθωθούν αναλόγως. Έπειτα η Γαλλίδα Υπουργό Περιβάλλοντος κυρία Σεγκολέν Ραγιάλ δέχτηκε να παραβρεθεί σε μια συνεδρίασή μας. Αναζητούμε μια κατάλληλη ημερομηνία. Ψάχνουμε να βρούμε μια, συμφων... μια ημερομηνία. Γι' αυτό και θέλω να ζητήσω κάποια ευελιξία από πλευρά σα, αν βρούμε κάποια έξτρα ημερομηνία είτε στο Στρασβούργο είτε στις Βρυξέλλες. Οι επαφές με υπολείπους υπουργούς συνεχίζονται. Έχετε σχόλια? That is not the case. Όχι. Οπότε... Μπορούμε λοιπόν τότε να προχωρήσουμε στην ακρόαση. Α, ναι. Συγγνώμη. Πάντα ξεχνάω να εξασφαλίσω ότι έχουμε συμφωνήσει για τα πρακτικά της συνεδρίασης της 12 η και 13ης Σεπτεμβρίου το 2016. Έχετε online στους φακέλους της Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, συγκρίνονται. Προχωράω τώρα στην ακρόαση του κυρίου Αντώνιο Εράριο. Καλωσορίσατε κύριε Εράριο. Είναι τμήματάρχης ε, του Τμήματος Διεθνή Ρυθμιστικά Ζητήματα του του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Ιταλίας. Σας ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και δεν θα κάνω άλλες εισαγωγικές παρατηρήσεις. Θα σας δώσω αμέσως το λόγο για να κάνετε τα δικά σας σχόλια για να ξεκινήσουμε μετά την ακρόαση. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μπορώ να μιλήσω Ιταλικά. Ναι, ωραία. σα ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Καταρχά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, την πρόεδρο τη Επιτροπή Έμει, ε, που με κάλεσε να συμμετέχω στη σημερινή συνεδρία. Είμαι ευτυχή που αντιπροσωπεύω εδώ τη Γενική ε, Διεύθυνση Οχημάτων που είναι μία από τι διευθύνσει του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που είναι η αρμόδια αρχή για την ε, πιστοποίηση των οχημάτων στην Ιταλία και είναι επίση η αρχή που συμμετέχει στι διεθνεί στους διεθνούς οργανισμούς όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τα οχήματα. Πρόκειται για μια, ένα δημόσιο οργανισμό που απασχολεί ε, στην πιστοποίηση γύρω στους 200 υπαλλήλους τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και στο περιφερειακό επίπεδο στα κέντρα έγκρισης ε, των ε, οχημάτων. Το θέμα των εκπομπών είναι πάρα πολύ σημαντικό και η έρευνα που κάνει αυτή η Επιτροπή είναι επίσης ε, πολύ σημαντική. Φάνηκε δε ότι τα οχήματα diesel πέρα από αυτά που παράγει η Volkswagen όπου είχαν τοποθετηθεί συστήματα ε, παράνομα. Ε, ακόμα λοιπόν και αυτά τα αυτοκίνητα τα οποία δεν φέρουν ε, τους, ε, τις συσκευές αυτές που έφεραν τα Volkswagen και είναι σύμμορφα με τους κανόνες. Πέρα από όλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες φορές εκπομπές οξυδίων ε, του αζότου πιο, πιο, σε πιο υψηλά επίπεδα από αυτά που είναι τα αποδεκτά και από, από αυτά που φαίνονται στις εργαστηριακές δοκιμές. Βλέπουμε λοιπόν ότι επιβάλλεται η τροποποίηση ε, συγκεκριμένων ε, μεθόδων ελέγχου όπως ας πούμε το σύστημα EGR και όλα αυτά σύμμορφα με τον κανονισμό 715 του 2017 ευρώ 5 και ευρώ 6. Θα πρέπει να σας πω και αυτή είναι και η άποψη του Ιταλικού Υπουργείου ότι όσον αφορά τα αριθμιστικά ζητήματα έχουν γίνει πολλά βήματα μπροστά τους τελευταίους μήνες. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις εκπομπές έχει εξελιχθεί έτσι ώστε να μπορούν να διευκρινιστούν οι μέθοδοι ελέγχου για να μπορούμε να ανταποκριθούμε και σε ελέγχους ε, υποσυνθήκες πραγματικής οδήγησης. Οι κατασκευαστές εντός του 2017 θα πρέπει να κάνουν ε, δοκιμές και σε κανονικές συνθήκες ε, οδήγησης στους δρόμους σύμφωνα με τον κανονισμό 2016-646 και θα πρέπει να καθορίσουν τις ε, διαδικασίες λειτουργίας καθώς και τις συμπληρωματικές στρατηγικές για τον έλεγχο των εκπομπών καθώς και τις στρατηγικές ε, για τον έλεγχο των εκπομπών. Πέρα από την πρόσφατη έγκριση από βουλευτές Κομισιόν μιας νέας διαδικασίας για τον έλεγχο στο εργαστήριο, τον ε, κύκλο WLTP, που είναι ένας, ένα παγκόσμιο πρότυπο για τον έλεγχο των ε, ε, οχημάτων, των εκπομπών των οχημάτων και τέλος ε, Εξετάζεται από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο ένας νέος κανονισμός πλαίσιο για την πιστοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που καλύπτει πάρα πολλά θέματα αλλά εγώ θέλω να τονίσω ότι ας πούμε το συγκεκριμένο σημείο είναι πολύ σημαντικό ότι δηλαδή θα μπορούν οι αρχές της πιστοποίησης να έχουν στη διάθεσή τους συγκεκριμένους μηχανισμούς ελέγχου, συσκευέ ελέγχου για να ελέγχουν τις πραγματικές εκπομπές των οχημάτων. Θεωρούμε λοιπόν ότι γίνονται πολύ σημαντικά βήματα μπροστά ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εκπομπές των οχημάτων θα είναι σύμφωνοι ε, θα είναι σύμφωνες με τις εκπομπές σε, πραγματικό, σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Και εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε. Επίσης, ευχόμαστε ότι θα είναι η δική μας συμβολή χρήσιμη για να διευκρινιστεί η, διευκρινιστούν οι πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος. Και πάλι σας ευχαριστώ για τη σημερινή πρόσκληση. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για αυτή σας την εισήγηση. Ξέχασα να αναφέρω ότι βέβαια όλοι οι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι πρόκειται για την πρώτη ακρόαση πολλών επομένων που τονίζουν το τι γίνεται στα κράτη-μέλη. Και εσείς είστε το πρώτος. Θα δώσω αμέσω το λόγο στον κύριο Σάλμπα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Ράριο. Η, προφανώς υπάρχει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά Εξίσου προφανώς θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ό,τι αφορά τις διάφορες ε, διαδικασίες έγκρισης τύπου στα διάφορα κράτη-μέλη. Δεδομένου ότι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, δικαιολογείται η διαφορά στην εφαρμογή της μεταξύ κρατών μελών, κατά την άποψή σας. <coughs> Σας ευχαριστώ. Όχι, ε, είναι ένας, ε, μια, η προδιαγραφή για την πιστοποίηση σε ολόκληρη την Ευρώπη από το 1990 και μετά έχουμε απόλυτα εναρμονισμένη διαδικασία πιστοποίηση. Και αυτό ισχύει για ολόκληρο το όχημα. Δεν είναι μόνο για τι εκπομπέ. Δεν περνάμε δηλαδή από ένα εθνικό καθεστώ στο ευρωπαϊκό. Αυτό ήδη ισχύει. Αυτό που είπα είναι ότι θα έχουμε περαιτέρω κανόνε που θα ε, συνδυαστούν με του υφιστάμενου κανόνε και θα μα επιτρέψουν ε, καλύτερα να μπορούμε να μετρήσουμε τι εκπομπέ και ε, στο δρόμο, δηλαδή να, να προσεγγίσουμε τις δοκιμές στην πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή οι δοκιμές γίνονται μόνο στο εργαστήριο δηλαδή και κυρίως βασίζονται σε μια διαδικασία ελέγχου που είναι μάλλον ξεπερασμένη. Οπότε κατά την άποψή σας, αν κατάλαβα καλά, δεν υφίστανται διαφορές στις ε, διαδικασίες έγκρισης τύπου μεταξύ των κρατών μελών. Δεν υπήρχαν τέτοιου είδους διαφορές κατά την άποψή σας. Όσον αφορά τι ε, εκπομπέ ε, που ρηπαίνουν σε περιορισμένο βαθμό, γιατί όπω σα είπα η προδιαγραφή είναι η ίδια. Πρόκειται για μια διαδικασία πιστοποίηση στο εργαστήριο, δηλαδή οι τεχνικοί ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πολύ καλά ε, καθορισμένο πρωτόκολλο. άρα λοιπόν το περιθώριο διαφορά ανάμεσα στην μια αρχή και στην άλλη δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Τώρα βέβαια όπως σας είπα ε, το τι συμβαίνει στο δρόμο σε πραγματικέ συνθήκε οδήγηση είναι που διαφέρει. Αλλά πάντω η πιστοποίηση, αν έχει γίνει στην Ιταλία ή στη Γερμανία, αυτό δεν πρέπει να έχει καμία διαφορά. Γιατί οι κανόνε είναι κοινοί. Επίσης είπατε ότι έχουν, έχει γίνει σημαντική προοδο Συμφωνώ, αλλά θα πρέπει να γίνει και άλλη πρόοδος. Ε, αν κατάλαβα καλά την άλλη μεριά, η Ιταλία επιθυμεί την ε, ε, αναβολή της θέσης σε ισχύ των νέων διαδικασιών έγκρισης τύπου. Για ποιο λόγο το επιθυμεί αυτό η Ιταλία. Κοιτάξτε, ίσω θα πρέπει κάπω να καθαρίσουμε το ερώτημα. Κοιτάξτε, η Ιταλία δεν έχει κάνει καμία πρόταση για αναδρομική ισχύ. Αν αναφέρεστε στην έναρξη ισχύω τη δοκιμή ε, ε, στο δρόμο, σε πραγματικέ συνθήκε. ναι. Εδώ απαντήσαμε σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα, δεν θυμάμαι τώρα το νούμερο, νομίζω είναι το νούμερο 9. Όχι, όχι, δεν είναι η 4, είναι η 5. Ε, Ερώτηση 5. Αν θέλετε γι' αυτό να μιλήσετε, να σας δώσω πληροφορίες. Έχουμε λάβει μέρος δραστήρια συνεργασία που οδήγησε στην έγκριση του πακέτου ε, Χρειάστηκε πολύ χρόνος, όχι, όχι όμως επειδή δεν συμφωνούσαμε, γιατί και η ίδια η Επιτροπή έπρεπε να αναπτύξει ένα πρωτόκολλο ελέγχου για κάποια δοκιμασία, την οποία, το οποίο μας υπέβαλε τους τελευταίους μήνες και κυρίως χρειάστηκε να επαληθεύσουμε και πρώτη-πρώτη κομισιόν ότι υπάρχουν εξοπλισμοί κατάλληλοι για να μπορούν να μετρούν στον δρόμο τις εκπομπές. Γιατί καλή βούληση από την πλευρά των αρχών υπήρχαν, αλλά πρέπει να έχουμε και φε, φε, και όχι βαριές συσκευέ, για να μπορούμε να κάνουμε ε, δοκιμές, όπως σα είπα, ε, αρκετά αξιόπιστες. Πρόκειται λοιπόν για εξοπλισμούς ε, ακριβούς που τώρα με το τεχνικό κύπρο πρόοδο έχουν τέτοιε διαστάσει που να μπορούν να υπάρχουν μέσα σε κάθε αυτοκίνητο αλλά να δίνουν και αξιόπιστα αποτελέσματα. Θα πρέπει να μπορούμε λοιπόν να μετρήσουμε και τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες καθώς και τα μεγέθη των σωματιδίων κτλ. Από την τεχνική πλευρά λοιπόν έχει γίνει πρόοδος, από την πλευρά όμως της ε, ε, κοινή βούληση φάνηκε ο πλευρά όλων των κρατών μελών ότι να εισαχθεί ένα έλεγχο σε μια δοκιμή RDA ε, που θα είναι δεσμευμένη με το χρονοδιάγραμμα του Euro 6 δεν ήταν εφικτό, γιατί το Euro 6 έχει ήδη εγκριθεί και μπήκε σε εφαρμογή το 14 2015 Έχουμε ήδη δηλαδή αυτοκίνητα Euro 6 τα οποία έχουν πιστοποιηθεί κανονικά. Το θέμα ήταν να ε, ξεκινήσει αυτή η δοκιμή RDA και επίσης τα αυτοκίνητα Euro 6 να μπορούν να δοκιμαστούν και στο δρόμο, σε πραγματικές συνθήκες. Θα είχαμε δηλαδή μια πρώτη φάση για εκμάθησης και για την ίδια την ε, αυτοκινητοβιομηχανία που θα έπρεπε να διαπιστώσει αν όντω είναι αξιόπιστες αυτές οι δοκιμές και για αυτό το λόγο η συζήτηση εστιάστηκε στον παράγοντα συμμόρφωσης, δηλαδή να προσπαθήσουμε να συσχετίσουμε τις εκπομπές στο εργαστήριο, που όπω ξέρουμε δεν είναι πολύ αντιπροσωπευτικέ, με τις εκπομπές ε, στον δρόμο. Εάν είχαμε διαλέξει ένα παράγοντα συμμόρφωσης ένα προς ένα, τότε κανένα όχημα δεν θα ήταν πια δυνατόν να πιστοποιηθεί από το 2017 και στο εξή. Γι' αυτό και η Κομισιόν αποφάσισε να φτιάξει ένα χρονοδιάγραμμα σε δύο φάσεις. Μια πρώτη φάση που ξεκινά το 2017, κάπως πιο αμβλία και δώσει γενική συζήτηση για τον παράγοντα συμμόρφωσης. Κάθε κράτος μέλος ενημερώθηκε από τους κατασκευαστές να δούνε ε, τι ε, είδους τεχνολογίες υπάρχουν και από την Ιταλική πλευρά, όπως και τα άλλα κρατημέλη, θέλαμε να έχουμε έναν παράγοντα στην αρχή 3, μετά 2, μετά 5 2,5 και να βρει, βρεθεί μια συμβιβαστική. Και έπειτα μιλήσαμε για ε, χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και στην Ιταλία δεχτήκαμε ένα συμβαστικό πακέτο που σίγουρα δεν το αποφασίσαμε εμείς, μας το πρότεινε η Κομισιόν, αλλά υπήρχε η στήριξη δύο μεγάλων κρατών μελών και γι' αυτό και καταλήξαμε σε μια συμβιβαστική που ήταν αποδεκτή ως πρώτη φάση. Διακόπτη η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Έχουμε πολλές ερωτήσεις, οπότε θα επανέλθουμε. Καλό είναι να απαντάτε ακριβώς στην ερώτηση, γιατί διαφορετικά παίρνει πολύ χρόνο η συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε μαζί μας ε, σήμερα που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Μου πρόκαλεσε κάπως έκπληξη το θετικό σχόλιο που κάνατε για την ε, το RTE και για την ε, εξέλιξη στην Ιταλία, γιατί η Ιταλία είναι η κατευθυντική χώρα που καθυστερεί τη διαδικασία αυτή. Από ότι φαίνεται από όλα τα έγγραφα της Τεχνικής ε, Επιτροπής. Μία άλλη ερώτηση έχω να σας κάνω. Στην ερώτηση 4 απαντήσατε. Με έναν ορισμό των απαγορευόμενων ε, συσκευών αναστολής όταν έχουμε σαφώς διαφορετική συμπεριφορά του οχήματος ε, στα εργαστήρια και στο δρόμο. Αυτό είναι λογικό. Αλλά στην ερώτηση 8 απαντάτε ως εξή. Αναφέρετε ότι ποτέ δεν ερευνάτε και δεν θα ερευνήσετε τις πραγματικές εκπομπές ε, στο δρόμο. Θα κάνετε μόνο έρευνες σε εργαστήριο. Άρα ποτέ δεν θα διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ του εργαστηρίου και του δρόμου. Ποτέ λοιπόν θα, θα ανακαλύψετε τέτοιες συσκευές αναστολής. Μα αυτό είναι το ονειρικό σενάριο των όσων θέλουν να παραβιάσουν τον νόμο. Σαν να λέει η αστυνομία, α, εμείς θα ελέγχουμε 9 με 5. Άρα οτιδήποτε εγκληματική δραστηριότητα από τι 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 το πρωί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εμείς δεν θα ελέγξουμε. Μπορείτε παρακαλώ να σχολιάσετε τα επικριτικά σχόλια αυτά. Ευχαριστώ. Αυτό που είπαμε, τώρα δεν θυμάμαι αν ε, είναι στην τέσσερα ή, κάτι άλλο, ή σε κάποια άλλη ερώτηση. Εμείς ως αρχή πιστοποίησης εφαρμόζουμε τον κανονισμό. Και ας πούμε ε, ότι μέχρι σήμερα, πριν από το RDE, η πιστοποίηση δίνεται με βάση συγκεκριμένο πρωτόκολλο και συνθήκες εργαστηρίου όμως. Πέρα από αυτές τις συνθήκες δεν έχουμε εμεί εξουσία για να πούμε στον κατασκευαστή κοιτάξτε ε, ότι εδώ ακολουθείται μια στρατηγική που δεν γίνεται δεκτή, δηλαδή εκτός του κύκλου. Εφαρμόζεται ο κύκλος της δοκιμής και αν το αποτέλεσμα είναι θετικό πιστοποιείται. Αν δεν είναι δεν πιστοποιείται. Αυτό έλεγα και στο συνάδελφό σας. Όλες οι αρχές με τον ίδιο τρόπο κινούνται Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Ναι, ναι, βέβαια, συγγνώμη που σα διακόπτω. Ε, γνωρίζατε όμω για τη χρήση αυτών των ε, μηχανισμών ε, μείωση τη ρήπανση στη διάρκεια των δοκιμών, των κύκλο δοκιμών. Το γνωρίζετε, ναι, αλλά αυτό είναι, υπάρχει, είναι γραμμένο σε πάρα πολλές μελέτες από το κοινό ερευνητικό κέντρο που θα έπρεπε να το γνωρίζετε. Προσπαθήσατε ποτέ να ελέγξετε κατά πόσο τα αυτοκίνητα ήταν πειραγμένα, όπως ε, είπε ο πρώην ε, Επίτροπος Ποτότσνικ, για να είναι σύμμορφα με το αυτό το τεστ στα εργαστήρια ε, και όχι στον δρόμο. Εσείς προσπαθήσατε να ελέγξετε τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Όχι. Δεν γνωρίζαμε την ύπαρξη τέτοιων μη αποδεκτών, μάλλον τη, τη χρήση τέτοιων μη αποδεκτών συστημάτων. Αρχίσαμε να το ερευνάμε ε, αμέσως μετά το ξέσπασμα αυτού του σκανδάλου της Volkswagen. Προηγούμενα δεν είχαμε ελέγξει, γιατί εμείς κάναμε τη δουλίτσα μας. Ελέγχαμε σύμφωνα με τις προδιαγραφές τα οχήματα στο εργαστήριο. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Μου αρκεί αυτό. Δεν το έχετε ελέγξει. Το άλλο ερώτημα που έχω να σας κάνω. Σε ό,τι αφορά τα 22 λεπτά, τα οποία χρειάζονται η Fiat για να θέσει εκτός λειτουργίας τη συσκευή. Δεν το παραμελείτε αυτό, αλλά αυτό πιστεύετε ότι είναι σύνομο, γιατί αποτελεί μια ρύθμιση για την προστασία της μηχανής, του κινητήρα. Αυτό αληθεύει αφενός. Και άλλη ερώτηση. Και κατά δεύτερον, αν ε, αυτή η συσκευή πρέπει να απονεργοποιηθεί μετά από 22 λεπτά. Υπάρχουν πολλά άλλα συστήματα τα οποία δεν χρειάζεται να απενεργοποιήσει μετά από 22 λεπτά. Άρα, γιατί συμφωνείτε με τη δήλωση αυτή, γιατί δίνετε πιστοποίηση τύπου όταν πολύ απλά δεν είναι σύμφωνα με τον νόμο. Il veicolo ha rispettato la normativa perché il laboratorio ammesso che il sistema si spenga. Eh, eh, Κοιτάξτε, κάθε άλλη αρχή που είχαμε ερωταπαντήσεις γραπτές, όλοι είπαν ότι αυτή η αλλαγή χρόνου ε, είναι ε, αυτή, αυτή αυτός ο διακόπτης χρόνου είναι η τέλεια ε, περίπτωση ενός τέτοιου μηχανισμού. Ναι, αυτό θα γινόταν όντως αλήθεια αν το σύστημα γινόταν να σβήσει. Αυτό το είπε η KBE που είναι η γερμανική αρχή πιστοποίησης. Εμείς δεν το επιβεβαιώσαμε αυτό και θα γνωρίζετε πως υπάρχει και μια επιτροπή διαμεσολάβησης για να συζητήσουμε τεχνικά το θέμα. Για να είμαι σύντομος, το σύστημα που υιοθέτησε ε, ε, η Fiat ε, δεν είναι ένα σύστημα το οποίο σβήνει, είναι ένα σύστημα το οποίο τοποθετείται σε ένα όχημα Euro 6 το οποίο έχει δύο κυκλώματα GR κυκλοφορίας δηλαδή. Το ένα χάνει τη λειτουργία του αλλά το άλλο συνεχίζει να λειτουργεί και η απόδειξη είναι ότι αν κάνεις αυτό το, το τεστ σε ένα όχημα θα έχεις ακόμα και αν το σβήσει, θα έχεις εκπομπές 13 φορές περισσότερο από τις επιτρεπόμενες όσον αφορά τα οξύδια του αζότου. Το σύστημα συνεχίζει να λειτουργεί και εντός των νομίμων ορίων κατά τη γνώμη μας. Όταν θα έχουμε βέβαια τις ε, δοκιμές στο δρόμο, όλα αυτά θα παίξουν όσον αφορά τη βελτίωση ε, των επιδόσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ θα σας κάνω τις ερωτήσεις στα γερμανικά. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τις απαντήσεις σας τις οποίες λάβαμε και γραφτά. Να αναφερθώ και στην ερώτηση του κ. Γκριμπράντη, η οποία είναι και πολύ ενδιαφέρουσα. Επειδή οι πληροφορίες αυτές κινούνται λίγο προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Μετά από 20 λεπτά λοιπόν, τι γίνεται ακριβώς στη Fiat ε, από, απενεργοποιείται και συσκευή, δεν απενεργοποιείται. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το άλλο ερώτημα είναι το εξή. Είπατε ότι μετά από 20 λεπτά α, η λειτουργία αυτή απενεργοποίηση έχει ω σκοπό την προστασία του κινητήρα. Μα τι θα πρέπει να προστατευτεί σε περίπτωση ανακυκλοφορία καυσαερίων. Δεν το καταλαβαίνω αυτό από τεχνική άποψη. Λοιπόν, Επιβεβαιώνω ότι το σύστημα δεν σβήνει, συνεχίζει να λειτουργεί, ακόμα και αν τροποποιηθεί, δηλαδή δεν λειτουργεί στο 100% αλλά το ένα από τα δύο κυκλώματα χάνει σε ένταση. Τι πρέπει να προστατεύσουμε κάποια συστατικά του συστήματος GR, ε, δηλαδή το σύστημα κυκλοφορίας ε, και εκπομπής των ε, ρήπων, γιατί σημαίνει ε, αυτό ότι μπορεί να μπλοκαριστεί, μπλοκαριστούν οι βαρβίδες του ECR και να οδηγηθούμε σε ατυχήματα πολύ σοβαρά. Γνωρίζουμε περίπτωση όπου μπλοκάρισε το EGR στον αυτοκινητόδρομο και άρα το, ο κινητήρας σβήνει αυτόματα, χωρίς καμία προειδοποίηση. Για να αποφύγουμε λοιπόν ε, τέτοιες αποθέσεις ε, ανθρακούχες ε, που δημιουργούνται από το EGR να αλλάσουν κάποια συγκεκριμένα τμήματα συστατικά είναι να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε με λιγότερη ένταση. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα ε, συμφωνείτε ή όχι τεχνικός και γι' αυτό και το συζητάμε. Και γι' αυτό και επαναλαμβάνω ότι με τον κανόνα RDE η διάρκεια θα εξελιχθεί. Γιατί δεν πρόκειται για δοκιμή στο εργαστήριο, αλλά για μία δοκιμή στον δρόμο που θα διαρκεί μάλιστα 90 λεπτά, από όσο γνωρίζω. Ευχαριστώ. Ναι, για το ερώτημα αυτό υπάρχει μία διαφορετική απόψη σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Οχημάτων θα γίνει σχετική ακρόαση αυτή την εβδομάδα και θα θεω ερευνήσουμε αυτό, γιατί από διατροτικής άποψη υπάρχει το εξή πρόβλημα. Αν υπάρχουν διαφορετικέ ερμηνείε από τι υπηρεσίε και έχουμε ένα ενιαίο κοινωτικό δίκαιο το οποίο όμω εφαρμόζεται διαφορετικά σε κάθε χώρα, πώ θα επιληθεί αυτή η διαφορά. Εσεί έχετε μια, κάποια άποψη σε ό,τι αφορά τις διαφορετικές αυτές ερμηνείε. έχετε επευθυνθεί προ την Κομισιόν, έχετε για παράδειγμα συνεργασία με το ΚΑΜΠΕ ή άλλες τέτοιες υπηρεσίες. Guardi, dopo oh, eh, il cosiddetto Dieselgate, noi abbiamo avuto delle... Κοιτάξτε, μετά από το Dieselgate, εμείς κάναμε συνεδριάσεις, ανάμεσα, επαφές ανάμεσα στις ε, αρχές επιστοποίησης, όπου μιλήσαμε για αυτές τις διαφορές ερμηνείας. Και μάλιστα Πήγαμε εμεί στο Βερολίνο, φιλοξενούμενοι του Γερμανικού Υπουργείου, την παρουσία του KBA της Γερμανίας και της ε, αρχής του Λουξεμβούργου και της Ολλανδίας και μάλιστα σε συμπεράσματα του Γερμανού συναδέλφου που έχουμε εμείς εδώ σε διαφάνειες λέει ότι υπάρχει αυτός ο κανόνας ε, after fallet. Δηλαδή, και εδώ αναφέρομαι στο, στις συσκευές ε, μείωσης. Γιατί έχουμε ένα σωρό, ένα κανονισμό που δέχεται αυτό τη συσκευή και έχουμε εκατοντάδες σελίδες εφαρμοστικές μετά και δεν γίνεται ούτε μία αναφορά στο άρθρο 5.2 του κανονισμού Euro 5 και Euro 6, το πρόβλημα εκεί έγκυται. Είναι αλήθεια μάλιστα ότι σε επίπεδο του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών που έγινε στις 7 Ιουνίου του 2016, πολλοί είπαν, υπουργοί είπαν στην Κομισιόν ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να αναπτυχθούν κατευθύνες γραμμές ώστε να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι είναι εντάξει και τι όχι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει ένα σταθερό σημείο και οι αρχές να γνωρίζουν ότι συγκεκριμένε τεχνικέ λύσει είναι εντάξει, άλλε όχι. Μέχρι στιγμή επικρατεί αυτή η αβεβαιότητα. Για μας δεν υπάρχει αβεβαιότητα, γιατί τη απουσία συγκεκριμένων κανονισμών αυτός, αυτή η συσκευή είναι πιστοποιήσιμη. Δηλαδή δεν πιστοποιούμε εμείς τη συσκευή, πιστοποιούμε το όχημα. Το όχημα περνάει την δοκιμή, τέλος της υπόθεσης, δίνουμε την πιστοποίηση. Ευχαριστώ. Στην ερώτηση 5 υπενθυμίζουμε το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διάφορες διαδικασίες επί παραβάση εναντίον της Ιταλίας ε, μεταξύ αυτών και το θέμα των ρήπων ε, οξυδίων του αζότου. Αυτό είναι ένα γεγονός. Όταν η Ιταλία αποφάσισε στη συνεδρία της CTVM τον Οκτώβρη ε, να ναι, να, να ζητήσει μια ε, αναβολή από το 2017 στο 2019 της ε, εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού ε, κύκλου οδήγησης. ποια ήταν η αντιδράσεις των συναδέλφων σας. το Υπουργείο Περιβάντος της Ιταλίας ε, συμφώνησε με, αυτή την, με αυτό το αίτημα ε, ή ήταν δική σας ε, πρωτοβουλία. Ah, guardi, fondamentalmente noi abbiamo... Βασικά, εμείς συνεργαζόμαστε με το περιβάλλον περιβάλλοντος, το, το Υπουργείο Βιομηχανίας και ούτω καθεξής. Αλλά αυτή είναι μια απόφαση που λήφθηκε από την Τεχνική Επιτροπή. Όπως έλεγα και πριν απαντώντας στον συναδελφό σας, ήταν μια τεχνική απόφαση γιατί διαπιστώσαμε ότι τα αυτοκίνητα Euro 6 είχαν κάποιους περιορισμούς και χρειάζονταν χρόνο για να προσαρμοστούν. Άρα λοιπόν, ε, αφού έγινε αυτή η επιλογή, ε, Εξετάσαμε την ε, βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, εξετάσαμε την προστασία του περιβάλλοντος, ήρθαμε και μάλιστα σε επαφή με άλλες χώρες που έχουν παρόμοια προβλήματα και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι όσο πιο γρήγορα ε, θα εγκρίναμε αυτό το πακέτο, τόσο πιο καλύτερα θα μπορούσαμε να εγγυηθούμε ότι θα είναι τουλάχιστον κάτω από συγκεκριμένα κατόφλια. Αλλά σίγουρα κατόλια. Ναι, συγγνώμη, διακόπτη. Συγγνώμη, αλλά πώ είναι δυνατόν να τηρήσετε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε ό,τι αφορά τι εκπομπέ και τα όρια εκπομπών των, του οξυδίων του αζότου και ταυτόχρονα ε, να εργάζεστε επί ενός ε, ευρωπαϊκού κύκλου που θα εφαρμοστεί όσο πιο αργά γίνεται. Ε, πώς ε, ε, συγκεράσονται οι, αποφ... οι απόψεις Υπουργείου Βιομηχανίας και Υπουργείου Περιβάλλοντος στην Ιταλία. Είναι πάντα συμβιβαστική αυτή η λύση. Εμείς δεν ζητήσαμε να αναβληθεί το 2019, μάλλον από το 2017 στο 2019. Όχι, η ημερομηνία του 2017 έχει παραμείνει. η προθεσμία για την καταγραφή όλων των αυτοκινήτων που ήταν για το 2018 ζητήσαμε να μετακινηθεί στο 2019 στο, πρόβλημα, στο πλαίσιο μιας συμβιβαστική λύσης. Γιατί όντως μέχρι, μέσα σε αυτήν την ε, Εντό αυτής μάλλον τη ημερομηνία θα έπρεπε να προσαρμοστούν όλα τα αυτοκίνητα. Μέσα στο πλαίσιο μιας συμβαστική, όπως σας είπα και στο ερώτημα 5, μπορούσαμε να έχουμε συγκεκριμένες και βέβαιες αξίες εκπομπών, ενώ σήμερα υπάρχουν υπερβάσεις για ορισμένα οχήματα κατά 450%. Εμείς έχουμε εθνικές εκθέσεις, ναι, έχω περιορισμένο χρόνο και θέλω να γνωρίζω για ποιο λόγο κάποιοι αυτοκίνητα στη διάρκεια της έρευνας στην Ιταλία ελέγχθηκαν από το Ινστιτούτο Μοτόρε του Εθνικού Ερευνητικού Κέντρου ε, και άλλα ελέγχθηκαν από το ιδιωτικό εργαστήριο του ομίλου FCA. Έχουμε σύμβαση με το Ινστιτούτο Μοτόρι της Νάπολης που είναι κρατικό Ινστιτούτο ανήκε στον Εθνικό Οργανισμό Έρευνας και εκεί ελέγχθηκαν και τέσσερα οχήματα της Fiat. Βέβαια, με, αφού λάβαμε τις πλήρες εκθέσεις, ε, θέλαμε να έχουμε μάλλον τις πλήρες εκθέσεις ε, εντός του Ιουλίου. Και νομίζω ότι η έκθεση αυτή φέρει μάλιστα την ημερομηνία της 27 Ιουλίου. Είναι ένα ερευνητικό εργαστήριο αλλά δεν έχει πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις, αποφασίσαμε να εμπλέξουμε και το κέντρο ελέγχου δοκιμών του Τωρίνου. Και εκεί το κέντρο δοκιμών του Τωρίνο βασίστηκε στα εργαστήρια FCA που είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα στάνταρ 17.000 της ΙΖΟ και είναι δυνατόν να παρακολουθήσει από πλευράς, ε, ή μάλλον για λογαριασμό του Υπουργείου, το εργαστήριο το ιδιωτικό. Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο ε, εργαστήριο δοκιμών. Εκεί μπορέσαμε να κάνουμε τις δοκιμές για ορισμένα οχήματα που διαφορετικά θα έπρεπε να γίνουν στην Νάπολη. Αλλά επειδή δεν είχαμε το χρόνο, έπρεπε να γίνουν όλες οι δοκιμές, ζητήσαμε από τους συναδέλφους του Τωρίνο να βοηθήσουν. Και γι' αυτό δουλέψαμε με δύο εργαστήρια. Δεν είναι σωστό να πείτε ότι έκανε τις δοκιμές η Fiat είναι κάτι που γίνεται τακτικά και από άλλε αρχές πιστοποίησης να χρησιμοποιηθούν οι εξοπλισμοί του κατασκευαστή, που είναι και εξοπλισμοί ενός συγκεκριμένου επίπεδου που έχουν μεγάλο κόστος. <laughs> sorry, sorry, late airplane. Ναι, συγγνώμη γιατί καθυστέρησε και το αεροπλάνο και καθυστέρησα και στις ερωτήσεις. Ε, σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ πέρα στην Επιτροπή εδώ πέρα προσπαθούμε να καταλήξουμε στο τι έχει ακριβώς συμβεί και τι μπορούμε να βελτιώσουμε στο μέλλον. Έχω μπει στην αίθουσα για την ανάγνωση των γράφων αυτών και από ό,τι φαίνεται η Ιταλία είναι από τα πιο ενεργά κρατημέλη σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Ουσιαστικά προσπαθεί να καθυστερήσει τη διαδικασία. Γιατί επειδή ως χώρα έχετε πληροφορίες τις οποίες πρέπει να μοιραστείτε μαζί μας για την τεχνική πρόοδο, για τις τεχνικές εξελίξεις. Γιατί βλέπουμε ότι, έχουν ότι υπάρχουν διαφορετικοί κατασκευαστές σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο και βλέπουμε ότι είναι πιο αυστηροί οι κατασκευαστές και η παραγωγή στην ε, στην Αμερική, στην Ασία, όταν μιλάμε για ένα καινούριο σύστημα, φαίνεται ότι η Ιταλία ήταν πολύ ενεργή στην καθυστέρηση της όλης διαδικασίας. Γιατί υπάρχει μήπως κάποια τεχνική πληροφορία που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας ή υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Νομίζω πως είχα απαντήσει στην αρχή της συζήτησης, αλλά επανέρχομαι θα, ε, ευχαρίστως. Αφού κάναμε την έρευνα για τα αυτοκίνητα EuroSafe, που πρόσφατα δηλαδή πιστοποιήθηκαν πριν από ένα ή δύο χρόνια, αποφασίσαμε, μάλλον και προτίσαμε, και προτείναμε και η Κομισιόν συμφωνούσε ε, ότι μέσα στη διαδικασία RDA η πρώτη τη φάση να είναι μια φάση όπου οι κατασκευαστές θα μπορούσαν να την περάσουν με προσαρμογές λογικές. Γιατί ένα προϊόν το οποίο μπήκε στην αγορά πριν δύο χρόνια δεν μπορεί να αλλάξει τελείως. Είναι επενδύσεις τεράστιες αυτές. Δεν έπρεπε να βρούμε μια συμβιβαστική για τα οχήματα πρόσφατης πιστοποίησης. Η Ιταλία λοιπόν έκανε τις έρευνές της και βρέθηκαν πιο ψηλές τιμές και μάλιστα οι δοκιμές που είχαν γίνει που πριν αναφέραμε στην Ιταλία και σε άλλες χώρες δείχνουν ότι ο παράγοντας συμμόρφωσης έξω από τον κύκλο είναι πολύ πάνω από το 3 και το 2,5. Άρα λοιπόν η επιλογή του 2,1 ως παράγοντα συμμόρφωσης είναι μια λογική επιλογή νομίζω ως πρώτη φάση. Να θυμίσουμε ότι Μόνο η Ευρώπη έχει την εμπειρία από την δοκιμή RDE. Ε. Δεν υπάρχουν παγκόσμια ε, τέτοιου τύπου δοκιμές, άρα δεν μπορούμε να πούμε. Να πούμε δηλαδή ότι μπορεί το αυτοκίνητο αυτό να λειτουργεί και να εκπέμπει κατά τον ίδιο τρόπο στη βουνό, στο λόφο, κοντά στη θάλασσα, στο ίσιωμα και γενικά. Εμείς θελήσαμε λοιπόν την πρώτη φάση να είναι λίγο πιο απαλή, αλλά η δεύτερη φάση πιο αυστηρή και νομίζω κάποιο το ανέφερε εδώ σε αυτό το ερωτηματολόγιο. Είχαμε ζητήσει παράγοντα συμμόρφωση 1,4. Ε, οι άλλε χώρε ζήτησαν περισσότερο και μάλιστα τελικά ε, καταλήξαμε στο 1,5 γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι το 2020 όταν θα αρχίσει να ισχύει πλήρως το πακέτο Θα έχουμε καταρχήν την ανοχή σφάλματος που και εκεί θα πρέπει να ορίσουμε το ποια θα είναι Εμείς δεν προσπαθούμε να καθυστερήσουμε τίποτα. Ίσως απλά να είμαστε πιο ρεαλιστές. Και δεχτήκαμε τη συμβιβαστική τελικά. Μάλιστα. Thank you. The is... Σας ευχαριστώ. Σημειώνουμε λοιπόν την απάντησή σας. Αυτό ήταν το σχόλιο που θα είχα να κάνω. Η θέση της Ιταλίας πάντως πιστεύετε ότι θα αλλάξει μετά την ε, ψηφοφορίας μετά τα όσα έγινε με το σκάνδαλο σε ό,τι αφορά την εκπομπή του διοξυβητού άνθρακα, των αζωτούχων, των νόξ. Ε, είναι όλα πολύ επιβλαβή για τις αστικές περιοχές και από ό,τι ξέρω και στην Ιταλία έχετε πάρα πολλές τέτοιες περιοχές όπου υπάρχει πυκνή ε, κυκλοφορία. Πιστεύετε λοιπόν ότι είναι κατεπήγον να υπάρχουν πιο αυστηροί κανόνες για να ανταποκριθούμε στα πρότυπα. Και κατά δεύτερον, τι νόημα έχει να θέτουμε πρότυπα και προδιαγραφές αν ουσιαστικά χρησιμοποιούνται συστήματα για να τα παρακάμψουν. Αν υπάρχει ένα παραθυράκι ε, σε ό,τι αφορά τα όρια εκπομπών για κάθε νομοθεσία. Ma guardi, noi abbiamo ε, sostenuto l'adozione del pacchetto RDE, l'adozione del nuovo ciclo ULTP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 Σημειώνουμε λοιπόν όσα σας είπατε και είναι καλό λοιπόν να εξετάσετε και εσείς ε, κάποιες από τις ε, ονοματοτήσεις όλων των εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι όλοι διατείνονται ότι τεχνικό πώς είναι εφικτό να περάσουν τα πρότυπα αυτά και να εφαρμοστούν σήμερα. Άρα νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να λυθεί υπόψη. Η κυρία Κίλιον. a very nice, nice name. Thank you. Uh, <clears throat> Χαίρομαι που είστε μαζί, μα είστε μαζί μας εδώ σήμερα. Δύο ερωτήσει έχω. Πρώτον, ε, συναντήσατε ε, να υπάρχουν, βρήκατε να υπάρχουν προγράμματα απόσυρσης αυτοκινητών στην Ιταλία. Ε, Ε, η Volkswagen ας πούμε έχει τέτοιου είδους ε, προγράμματα αν χρειαστεί κάποια επισκευή αυτή είναι η αν χρειαστούν κάποια επισκευή αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση Ευχαριστώ. Όσον αφορά την Volkswagen, στην Ιταλία υπάρχουν περίπου 750.000 αυτοκίνητα που πρέπει να ανακληθούν. Έχουμε πληροφορίες ε, βεβαίως από την Γερμανική Αρχή Πιστοποίησης, την KBA, ότι σταδιακά ε, κρίνει τις τεχνικού τύπου ανακλήσεις ανά είδος αυτοκινήτου, ανά μοντέλο αυτοκινήτου και έπειτα ο κατασκευαστής ε, από τον αντιπρόσωπο μάλλον στην Ιταλία, θα, θα δούμε και θα λαμβάνουμε τις πληροφορίες σε σχέση με την εκστατεία απόσυρσης αυτών των αυτοκινήτων. Όπως σας είπα, υπάρχουν και 7 οχήματα του ομίλου Volkswagen που αυτή τη στιγμή είναι στη διάθεση των δικαστικών αρχών, γιατί υπάρχει μία δικαστική διαδικασία στην Ιταλία και από αυτά τα οχήματα θα κάνουμε δοκιμές πριν να αποσυρθούν και μετά που θα έχει γίνει η απόσυρση, θα έχει μάλλον γίνει η ανάκληση των μοντέλων, γιατί θέλουμε να καταλάβουμε γιατί και πώς ακριβώς είναι η Και Φυσικά και δεχόμαστε τις δηλώσεις της ε, KBA, της Γερμανικής Αρχής, η οποία περιορίστηκε στο να μας πει ότι το αυτοκίνητο από τη στιγμή που θα έχει ανακληθεί θα είναι σύμμορφο προς την πιστοποίηση, όσον αφορά τις εκπομπές, όσον αφορά την υποδύναμη, την κατανάλωση, τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κτλ. Να όμως να δώσουμε απαντήσει στους καταναλωτές μας εμείς, γιατί δεν καταλαβαίνουμε τότε, αφού τα καταφέρνουν να είναι πιστοποιημένα και χωρίς αυτή τη συσκευή, δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο έγινε αυτό. Και θέλουμε να δώσουμε εξηγήσει λοιπόν και στου καταναλωτέ μα και κάνουμε τέτοιου είδου έρευνα. Ζητήσαμε πληροφορίε και από την KBA τη Γερμανία. Δεν έχουμε λάβει όλε τι λεπτομέρειε, αλλά εντάξει. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να το προχωρήσουμε και μόνοι μας. Ευχαριστώ. Από ό,τι ακούω, ε, δεν θέλετε να κάνετε δοκιμές σε, σε δρόμους, σε πραγματικές συνθήκες. Πώς θα αξιολογήσετε, πώς θα μετρήσετε την ε, επιτυχία του προγράμματος ανάκλησης αν δεν μπορείτε να κάνετε μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες. Allora, intanto parliamo... Καταρχάς, μιλάμε, ας μιλήσουμε για τα αυτοκίνητα της Volkswagen. Ωραία, ο κατασκευαστής έχει τοποθετήσει αυτή τη συσκευή, την παράνομη και το δέχτηκε και το KBA ε, όπως σας είπα, έχουμε κάνει δοκιμές στο εργαστήριο, αλλά θα κάνουμε και για το στο δρόμο. Θα γίνουν και δοκιμές στο δρόμο, γιατί θέλουμε να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του οχήματο. Βεβαίω, όμως, η δοκιμή στον δρόμο μας βοηθά να καταλάβουμε και το φαινόμενο. Γιατί ε, μέχρι στιγμή δεν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την πιστοποίηση μας. Ε, βοηθά στο να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του οχήματο. Ε, ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θέλω να περάσω στην ερώτηση 8 και μάλιστα συγκεκριμένη απάντηση σας λέτε ότι δεν είναι νομικά δυνατό να γίνουν εναλλακτικές ε, δοκιμές πέραν του NEDC. Ε, πού η νομοθεσία απαγορεύει τη χρήση τέτοιων άλλων εναλλακτικών δοκιμών. Μπορείτε να μου πείτε σε ποιο άρθρο. Όχι, δεν νομίζω ότι απαγορεύει κάποιο άρθρο. Όχι. κανόνας λέει ότι ένα εργαστήριο δοκιμών κάνει, εφαρμόζει το συγκεκριμένο πρωτόκολλο για τη συγκεκριμένη δοκιμή και δίνει την πιστοποίηση ή όχι. Εάν δούμε τον κανονισμό RDA, το τελευταίο δηλαδή που δημοσιεύθηκε, στο προήμιο υπάρχει ένα εκτιμώντας που η Κομισιόν το πρότεινε και το εκνέκριναμε κι εμείς, όπου γίνεται σαφώς αναφορά στην απουσία δοκιμής στο δρόμο. ώστε το αυτοκίνητο να μπορεί να, να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες χρήσης. Ε, το κανονισμός 715 του 2007 ε, λέει ότι πρέπει να γίνεται η δοκιμή στο εργαστήριο κτλ. Ε, αλλά αν υπάρχει ένα, μια δοκιμή, εφόσον προβλέπεται μια δοκιμή, δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε έλεγχος. Χρειάζεται πάντα να υπάρχει ένα τεστ αναφοράς, ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Τώρα θα υπάρχει αυτό και θα μπορούμε να πούμε ναι, αυτές είναι οι κανονικές συνθήκες και ανταποκρίνεται σε αυτό. Ωραία, χαίρομαι που λέτε ότι η νομοθεσία δεν το απαγορεύει ρητά, γιατί στην ερώτηση 10 αναφέρεται στην απάντησή σας ότι κάνετε πρόσθετες δοκιμές ε, και στον δρόμο. Τι άλλαξε η νομοθεσία, ε, πώς είναι τώρα δυνατόν να επιτρέπετε να κάνετε 14 διαφορετικές δοκιμές στον δρόμο. Ε, δοκιμές στον δρόμο δεν μας το ζήτησε κανείς. Αυτό είναι η πρωτοβουλία το Υπουργείο της Ιταλίας που δεν το κάνατε αυτό δηλαδή παλιότερα. Γιατί το σκάνδαλο της Volkswagen ξέσπασε το Σεπτέμβριο του 2015 και η Γερμανία, η Αγγλία, η, η, η Ολλανδία ξεκίνησαν τέτοιες δοκιμές. Εσείς δεν είχατε ποτέ αυτή την αίσθηση ότι καλό θα ήταν να κάνετε και πρόσθετες δοκιμές που κάνετε τώρα. Ενώ λέτε ότι προηγουμένως δεν σας επιτρεπόταν να κάνετε τέτοιου είδους δοκιμές. Κοιτάξτε, ε, τις επιπλέον δοκιμές δεν τις έκαναν οι ε, αρχές επιστοποίησης, τα τις, τις έκαναν ε, ερευνητικά κέντρα όπως το ICCCT ή το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο του Ίσπρα. Δηλαδή κάνουν διαφορετικά δουλειά από, διαφορετική δουλειά από ότι η αρχή επιστοποίησης. Έπειτα αρχη επιστοποιησης επειτα αυτες οι πληροφορίες οι αρνητικές μας ήρθαν, αλλά όχι τόσο που να μας κάνουν ε, να σκεφτούμε ότι αυτό έγινε με στόχο, αυτό έγινε με στόχο απάτη όπως για την Volkswagen. Το γνωρίζαμε γιατί η Κομισιόν μας είχε ενημερώσει και είχαμε ξεκινήσει να δουλεύουμε για την δοκιμή RDE που επιταχύθηκε. Ε, τώρα βλέπω ότι προβαίνεται σε πρόσθετες δοκιμές, πάλι καλά, λίγο καθυστερημένα. Ε, ελπίζω όμως ότι τώρα θα εξετάσετε και τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών, τώρα που γνωρίζετε τα πάντα πια. Και είναι ενδιαφέρον διότι έχετε κάποια αποτελέσματα που στην ίδια τη δική σας την έρευνα αυτοκίνητα εκπέμπουν περισσότερα ε, με ε, θερμή εκκίνηση από ότι με ψυχρή εκκίνηση. Ε, ζητήσαμε, ρωτήσαμε πολλούς εμπειρογνώμονες και μας είπαν ότι δεν υπάρχει λογική εξήγηση γι' αυτό. Ε, αυτός ε, ήταν μάλιστα και ο λόγος που η EPA προχώρησε σε βάθος στην έρευνα για τη Volkswagen. Υπάρχουν λοιπόν πολλά θέματα. Τώρα τα ίδια θέματα τα βρίσκεται ξανά και πάλι συμπεραίνεται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Πώς είναι δυνατό αυτό. Έχω την εντύπωση ότι κοιμόσασταν πριν και κοιμάστε και τώρα. <laughs> Όχι, δεν κοιμόμαστε. Δεν κοιμόμαστε, ξυπνήσαμε. Είμαστε πολύ ξύπνοι, ειδικά σήμερα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, εφαρμόζουμε του κανόνε. Το, το έχουμε σημειώσει και εμεί στην έκθεσή μα. Αν και ξεκινά κανεί ε, εν θερμό, είναι διαφορετική συμπεριφορά. Και αν ξεκινά κανεί εν ψυχρό, είναι διαφορετική συμπεριφορά. Αν όμω ξεκινάμε εν ψυχρό, έχουμε τώρα γίνεται η δοκιμή στο εργαστήριο Κοιτάξτε, δεν κάνετε μόνο την έγκριση τύπου, πρέπει να εφαρμόσετε και την νομοθεσία λόγω της οποίας απαγορεύονται οι μηχανισμοί ε, Δεν μιλάω για έγκριση τύπου, μιλάω για συμμόρφωση και εφαρμογή του νόμου. Guardi, eh, noi Κοιτάξτε, εμείς κάναμε τις δοκιμές μας με στόχο να ε, παληθεύσουμε αν υπήρχαν απαγορευμένοι μηχανισμοί αναστολής. Πέρα από τα Volkswagen, γιατί το είχαν τοποθετήσει οι κατασκευαστές, στην Ιταλία δεν βρήκαμε τουλάχιστον σε άλλα αυτοκίνητα ούτε και σε άλλες χώρες από όσο γνωρίζω. Η συμπεριφορά είναι κάπως παράξενη, γιατί πέρα από το κύκλο πιστοποίησης βγαίνουν οι εκπομπές. Αν όμως οι κατασκευαστές έχουν ε, φτιάξει ε, τους κινητήρες τους για να ξεπεράσουν αυτόν τον κανόνα, ίσως είναι πρόβλημα και το κανόνα που πρέπει να αλλάξει, να βγει από τον κύκλο, όπως το έκανε και το RTF. Εφόσον ε, ο κανονισμός λοιπόν βασίζεται σε ένα κύκλο που αναπτύχθηκε στα τέλη του 70 αρχές του 80, που ήταν απλώς τη σύγκριση, σύγκριση κάποιων οχημάτων, οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Όσοι ασχολούνται με την ποιότητα του αέρα θέλει Θέλουν αποτελέσματα, συγκεκριμένα, πραγματικά, πάντα. Αυτή η δοκιμή, αυτό το τεστ δεν είναι πια κατάλληλο. Γι' αυτό χρειάζεται το RDA, αλλά και το κύκλος WLTP. Είναι, όποιος δει λίγο το διάγραμμα θα δει ότι είναι πολύ πιο δυναμικό, αλλά χρειάζονται χρόνια για να υπάρξει μια τέτοια κοινή, ε, ένα κοινό πρωτόκολλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να επανέλθω στην απόφαση για το πού δοκιμάζονται τα οχήματα στην έκθεση που μας έδωσε το Υπουργείο Μεταφορών και ιδιαίτερα σε βάση αυτό που μας είπατε προηγουμένως. Θέλω να καταλάβω, ε, δεν νομίζετε ότι ήταν άστοχο το ότι χρησιμοποιήθηκαν εγκαταστάσεις ε, εντός του ομίλου Fiat, του ομίλου FCA. Ποιος έλαβε αυτή την απόφαση. Με λίγα λόγια. Ευχαριστώ. Το να χρησιμοποιείτε το εργαστήριο του κατασκευαστή και βεβαίω εντάξει, εσεί έχετε την άποψή σα και τη σέβομαι, όμω εμεί ω δραστηριότητα πιστοποίηση χρησιμοποιούμε τι εγκαταστάσει τη ΦΙΑ του Σωτορίνου εδώ και χρόνια και βασιζόμαστε στα εργαστήρια της Fiat. Γιατί όσο κάνουμε εμείς ε, μια δοκιμή σε ένα ε, γκαράζ, ε, γίνεται δοκιμή ταυτόχρονα και σε άλλο, για άλλο όχημα ας πούμε. Είναι συγκεκριμένα εργαστήρια ε, τα οποία είναι ανεξάρτητα αλλά τα λειτουργούμε εμείς εκείνη την ώρα μας δίνεται ο χώρος, το εργαστήριο. Και το Υπουργείο το γνωρίζει αυτό. Εδώ και χρόνια γίνεται αυτό. Το γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά. Άρα λοιπόν να σημειώσουμε ότι και τα ε, συγκεκριμένα εργαστήρια είναι λιγοστά λοιπόν. Μάλιστα ερώτηση 11, σε σχέση με την απουσία δοκιμών που γίνονται σε, για τρία οχήματα της ε, FCA, της Fiat. Γιατί αυτά τα τρία οχήματα φαίνονται στις πρώτες δοκιμές ελέγχου των κύκλων ψυχρό και θερμό και μετά δεν εμφανίζονται σε άλλες δοκιμές όπως έγινε για τα υπόλοιπα οχήματα. Και μάλιστα εξαφανίζονται εκείνα τα τρία με τις μεγαλύτερες εκπομπές οξυδίων του αζότου. Κοιτάξτε, είναι τα αέρο 5Β αυτά που λέτε. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 δεν μπορούν πλέον να κυκλοφορήσουν. Ε, για να εντοπίσουμε αυτά τα τρία οχήματα λοιπόν είχαμε κάποιες επιπλέον δυσκολίες. Μας, είχαν δοθεί, μας είχε δοθεί όμως μια προθεσμία για τις 27 Ιουλίου, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να δημοσιευθεί αυτή η έκθεση και γι' αυτό και ορισμένες δοκιμές δεν έγιναν. Αλλά το γνωρίζουμε, μπορούμε και να κάνουμε αυτές τις δοκιμές και μετά. Θα γίνει μάλιστα κάποιο αντέντομο σε αυτή την έκθεση, γιατί υπάρχουν διάφορα σφάλματα εδώ, τυπογραφικά και άλλα. Με ρωτήσατε γιατί λείπουν κάποιοι ρήποι. Για κάποιους ρήπους εδώ δεν το, δεν το γράψαμε γιατί είχαμε εστιάσει στο οξύδιο του αζότου. Έχουμε όμως τα στοιχεία η συμπεριφορά η ποιοτική αυτών των οχημάτων συμπεριλαμβανομένων των τριών της Fiat είναι γνωστή. Λείπουν κάποιες δοκιμές αλλά αυτό δεν θα προσθέσει τίποτα και κάποιος μάλιστα το έγραψε στον τύπο και αυτό με χαροποίησε ως Ιταλό γιατί και αυτό τα αυτοκίνητα και αυτό ακόμα τα οποία τα πήγαν χειρότερα είναι οχήματα τα οποία είναι της ε, Fiat Κανένα δεν μπορεί να πει ότι εμείς ε, παραχαράξαμε τα αποτελέσματα. Είναι τις ίδιες τη Fiat αυτά τα τρία οχήματα τα οποία ρηπαίνουν περισσότερο. Δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως παράληψη δηλαδή στις ε, δοκιμές μας. Κοιτάξτε, εδώ δεν προσπαθούμε να βρούμε μέσο όρο με βάση διαφορετικές αναλύσεις. Θέλουμε συγκεκριμένες αναλύσεις των μεμονωμένων ε, μοντέλων. Θέλω να καταλάβω καλύτερα γιατί αυτά τα τεστ σύγκρισης οχημάτων της Fiat με άλλα έγιναν και μάλιστα με κάποια οχήματα Fiat χρησιμοποιήσατε κύκλους Energy and Thermo ενώ για άλλα οχήματα χρησιμοποιήσατε τον κύκλο Urban και Artemis και μάλιστα για το Artemis μιλήσαμε πολύ εδώ στην Επιτροπή. Μπορείτε να μας πείτε πιο ξεκάθαρα ή να περιμένουμε να δούμε την έκθεση που ελπίζουμε να έρθει σύντομα. Ναι, να ξεκινήσω από την τελευταία σας ερώτηση δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί, δηλαδή δεν μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση, γιατί ακριβώς πρέπει να συμπληρώσουμε τις δοκιμές για τη Volkswagen. Να θυμίσω ότι είναι κομμάτια αυτή τη έκθεσης. Δεύτερον, Έχουμε διαβιβάσει την έκθεση στην Επιτροπή ΕΜΙΣ και εν να αυτήν εδώ της ακρόση γιατί ο Υπουργός ε, ζήτησε να ενημερωθεί η Πρόεδρος και η Επιτροπή σας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή είναι ακόμα ε, περιορισμένες Περιμένουμε ώστε να το ελέγξουμε, να το συμπληρώσουμε και να το συζητήσουμε και με το Ινστιτούτο των Οχημάτων ε, χρησιμοποιήθηκε ο κύκλος Urban γιατί θέλαν να δουν εκείνοι πώς συμπεριφέρεται το αυτοκίνητο σε ένα πιο δυναμικό κύκλο, δηλαδή σε αστικό περιβάλλον. Δεν έχει γίνει ωστόσο καμία παράληψη γιατί ο στόχος μας ήταν να αναζητήσουμε ε, μηχανισμούς αναστολής δεν βρήκαμε. Έπειτα, η ποιοτική συμπεριφορά συμφωνεί με τα όσα βρήκαν και άλλες χώρες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ. Στα γερμανικά. Καθηγητά Ράδιο. Κάποιες ερωτήσεις να σας κάνω. Στην απάντησή σας στην ερώτηση παριθμών 4 σχολιάζετε και τις κατηγορίες ε, της γερμανικής υπηρεσίας οχημάτων σε ό,τι αφορά κάποια μοντέλα της Fiat. Και επειδή καθυστερήσατε το αεροπλάνο μου, δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει ήδη το θέμα αυτό, αλλά προέκυψε ότι στη Fiat ε, η συσκευή αυτή απενεργοποιείται 22 λεπτά μετά την ε, θέση σε λειτουργία, δηλαδή περιέργως πώς, 2 ε, λεπτά μετά από την ε, περίοδο που προβλέπεται από τις εργοστηριακές δοκιμές. Είναι σύμπτωση. Ευχαριστώ. Το σύστημα δεν σβήνει, όπως είπα στο συναδέλφο σας. Τροποποιείται. Αποτελείται από δύο κυκλώματα και όχι ένα γιατί είναι όχημα Euro 6 όπου είναι πιο αυστηρό το όριο και χρειάζονται δύο κυκλώματα. Τουλάχιστον αυτή είναι η λύση που βρήκε η Fiat. Στα ένα από τα δύο κυκλώματα υπάρχει μία, ε, όπως είπα, σβήνει το ένα κύκλωμα και άρα υπάρχει μία ε, μείωση λειτουργίας. Γιατί διαφορετικά μπορεί να υπήρχαν βλάβες λόγω ε, αποθέσεων άνθρακα σε ευχαριστώ. Το κατάλαβα. Το αποδέχομαι. Και πού, από πού γνωρίζετε ότι απενεργοποιείται για την προστασία του κινητήρα. Γιατί το ρωτήσαμε τους ε, κατασκευαστές. Ζητήσαμε όλα τα software που είναι εγκατεστημένα σε αυτό το αυτοκίνητο. Έχουμε κάνει ελέγχους, έχουμε κάνει δοκιμές καταφέρατε να αποκωδικοποιήσετε και το λογισμικό. Sie die Software entschlüsseln? Το λογισμικό το αποκωδικοποιήσατε ή βασιστήκατε σε αυτά σωστά έδωσε ο κατασκευαστή. όχι, δεν φτάνουμε εμεί σε αυτό το επίπεδο. Εμεί κάνουμε δοκιμέ όπου είδαμε ότι το σύστημα μειώνεται και οι, οι τιμές των οξυδίων του αζότου αυξάνονται, αλλά δεν φτάνουν ποτέ στην τιμή 13 φορές παραπάνω που υποθέτει η γερμανική αρχή, που είναι η τιμή στην οποία φτάνει όταν σβήνει το σύστημα. Δεν σβήνει το σύστημα, όπως σας είπα, συνεχίζει να λειτουργεί. Είναι στο 6. Είναι, είναι μια μέτρια τιμή. Δεν είναι και χαμηλή, αλλά είναι μια τιμή στην οποία φτάνουν και, άλλες, και άλλα αυτοκίνητα. Στην ερώτηση 4, στην απάντησή σας, αναφέρετε ότι η υπηρεσία σας καλεί το γερμανικό, τη γερμανική υπηρεσία οχημάτων να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με αυτό. Αλλά η υπηρεσία σα θεώρησε ότι η περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Fiat και τη γερμανική υπηρεσία οχημάτων δεν ήταν απαραίτητη. Το γεγονό ότι σε εθνικό επίπεδο οι εθνικέ υπηρεσίε πιστοποίηση ερμηνεύουν το κινητικό δίκαιο ε, διαφορετικά θα έπρεπε να δικαιολογεί το γεγονό ότι η γερμανική υπηρεσία θέλει να έρθει σε επαφή με τη Fiat. Δεν πιστεύετε. Ε, νομίζω ότι υπάρχει εδώ μια παρεξήγηση. Κοιτάξτε, εμείς ε, διαμαρτυρηθήκαμε στη γερμανική αρχή γιατί καταλήγαμε ε, τέταρτη ή πέμπτη φορά να καλείται η Fiat στο Βερολίνο, Βερολίνο για να συζητήσει με την ε, KBA και δεν μας λέγανε, δίναν καμιά πληροφορία. Και στη Γαλλία υπήρξε μια επιτροπή έρευνα. Αλλά οι γαλλικέ αρχέ μα ζήτησαν από εμά όλε τι πληροφορίε σε σχέση με την πιστοποίηση του εν λόγω αυτοκινήτου. Ενώ η γερμανική αρχή δεν το έκανε αυτό. Μετά κάποια στιγμή τους, ε, στείλ, τους ενστήλαμε γιατί γνωρίζα, ε, μάθαμε τι γινόταν και παρακολου, τους παρακαλέσαμε να έρθουν σε επαφή μαζί μας, να μας πούνε τι τρέχει. Και αυτό μάλιστα προβλέπεται και από τους ε, κανόνες πιστοποίησης. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση. Τι μερίδιο έχει η Ιταλική κυβέρνηση, το Ιταλικό κράτος στην εταιρεία Fiat. Um, Δεν είμαι δικός. Δεν έχει μερίδιο το Ιταλικό κράτος. Είναι ιδιωτική εταιρεία ιδιωτικός όμιλος η ΦΙΕΤ. Δεν συμμετέχει το κράτος. We move now to the Και τώρα να περάσουμε στο δεύτερο γύρο της ακροασής μας και στρέφομαι προς τους συναδέλφους, τους έχω σημειώσει και τους δύο στον κατάλογο των ομιλητών. Εντάξει, πολύ ωραία. Και μετά έχω άλλα τρία άτομα στον κατάλογο, εκτός μικροφώνου όμως ομιλητής να σας ευχαριστήσω, Πρόεδρε, για τα χρονομιλία που μου δίνετε ακόμα. Να σας πω ότι η συνάδελφος Σαλίνη προφανώς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μιλήσει και να ρωτήσει διάφορα στοιχεία προ τον προσκεκλημένο μα, αλλά είναι στο αεροπλάνο, έχει καθυστερήσει και δυστυχώ θα χρησιμοποιήσω εγώ το χρόνο του. είναι το πρόβλημα αυτό τη Δευτέρα το πρωί. Αλλά θα ήθελα στα πλαίσια της γερμανοϊταλικής φιλίας να θέσω και την εξή ερώτηση σε σχέση και με αυτά που είπε η κυρία Εύη σε ό,τι αφορά την ερώτηση παριθμών 11. Και αναφέρατε ότι δεν υπήρχε ουσιαστικός λόγος να εξαιρεθούν από τους δοκιμές και από τους ελέγχους κάποια οχήματα. Η Αλφα Ρωμαίο, η Λάντσια, κάποιοι τύποι οχημάτων ελέγχονται ενδεχομένω διαφορετικά. Δεν σα κατηγορώ, αλλά θέλω να καταλάβω βάσει ποιων κριτηρίων κάνετε επιλογή των οχημάτων. Ε, eh, σα ευχαριστώ. Στην αρχή της ανάλυσης των δοκιμών σας έκανα μία ε, παρουσίαση για το ποια αυτοκίνητα κυκλοφορούν, τουλάχιστον τα Euro 5 και εκτός του ομίλου Volkswagen έχουμε καλύψει το 75% των αυτοκινήτων ε, Euro 5 ε, Β, αυτοκίνητα diesel που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην Ιταλία. Και αυτό για να είμαστε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικοί. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και θελήσαμε βεβαίω και να περιορίσουμε το κόστος, γιατί δεν είναι διόλο μελιτέο το κόστος όλων αυτών. Και μάλιστα να έχουμε αποτελέσματα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτά ήταν τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιήσαμε. Τώρα, για να επανέλθω στο γεγονός ότι ορισμένες δοκιμές παραλήφθηκαν, επαναλαμβάνω, αν υπάρξει δυνατότητα, που πράγμα που πιστεύω ότι θα γίνει, θα καταστεί ακόμη πιο ομοιογενής η, έκθεσή μας και καταλαβαίνω την, το ότι ρωτάστε γιατί σε ένα όχημα έγινε αυτή η δοκιμή και στο άλλο όχι. Αλλά πέρα από την δοκιμή εργαστηρίου που γίνεται υπό στάνταρ συνθήκες, όλες οι άλλες δοκιμές δεν μπορούν καν να είναι συγκρίσιμες. Δηλαδή, αν κάνουμε ε, στην Νάπολη για ένα συγκεκριμένο μοντέλο σήμερα ή και για ένα άλλο αύριο δεν είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα και μπορεί τη μια μέρα να κάνει ζέστη, την άλλη μέρα να κάνει κρύο κτλ. Στόχος είναι να, όπως είπα, σε αυτές τις δοκιμές ήταν να δούμε αν υπήρχαν εγκατεστημένες συσκευές αναστολής ή όχι και να δούμε κατά πόσο συμφωνήσαμε με τα όσα βρήκανε τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Το τι λείπουν αυτές οι τρεις δοκιμές για αυτά τα τρία οχήματα, όπως ε, κατά τύχη ε, είδαμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά αυτό δεν αλλάζει καθόλου τα αποτελέσματα της έρευνας και ε, το σκοπό αυτών των δοκιμών. Δεν θέλουμε να δούμε αν είναι σύμμορφα ή όχι τα οχήματα. Όλα τα οχήματα είναι σύμμορφα με τους κανονισμούς ε, στο εργαστήριο. Το θέμα είναι πώς συμπεριφέρονται στις πραγματικές συνθήκες και αν φέρουν ή όχι παράνομους μηχανισμούς αναστολής. Σας ευχαριστώ. Δηλαδή, αν μιλάμε για 75% ε, των οχημάτων diesel, ε, δεν θα, θα θεωρήσουμε ότι είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα και ότι δεν εξαιρέθηκαν κάποια συγκεκριμένα οχήματα. Σε ό,τι αφορά τώρα την ερώτηση που, που επικρίνεται την Γερμανική Υπηρεσία Οχημάτων, ε, για ελλείμματα στις απαντήσεις σας. Ε, μιλήσατε και εσείς για κάποια αντέντουμ, για κάποια πρόσθετα τα οποία θα δημοσιευθούν. Εγώ έχω να θέσω και κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, κοιτώντας την απάντηση υπαριθμών 2 στην επίσημη έρευνα. Εκεί ουσιαστικά δημοσιεύεται μόνο μία σύνοψη. Δεν δημοσιεύεται το σύνολο της έρευνας. Έχετε κάτι να κρύψετε. ή μήπω θα δημοσιεύσετε για σκοπού διαφάνεια στο σύνολο τη Έκθεση. Ε, Μάλιστα, ευχαριστώ. Όχι, δεν έχουμε κρύψει τίποτα. Όλα τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας έχουν δημοσιευθεί. Βεβαίως, ορισμένες τιμές εκπομπών, πέρα από τα οξύδια του αζότου, ας πούμε για τα μικροσωματίδια, τα έχουμε, αλλά δεν τα έχουμε δημοσιεύσει, γιατί η προσπάθεια των, για τις δοκιμές είχε στόχο τα οξύδια του αζότου και κατά πόσο ή όχι υπήρχε συσκευή αναστολής επαναλαμβάνω, και με το εργαστήριο της Νάπολη Έχουμε δημοσιεύσει γιατί κάποιες πληροφορίες από αυτές μπορεί να είναι ενδιαφέρουσες για όποιον κάνει έρευνες και η Κομισιόν μας ζήτησε κάποιες παραπάνω πληροφορίες. Να σας διακόψω όμως ε, λίγο γιατί δεν έχω έξι λεπτά. Το ερώτημα είναι το εξής. Στην απάντηση μόνο δύο λέτε. Αποφασίστηκε να δημοσιευτεί μόνο η σύνοψη, η σύνοψη μόνον. Εδώ προτίθεστε να δημοσιεύσετε το σύνολο της έρευνας. Η έκθεση θα μείνει ε, αυτή, γιατί ήταν απόφαση εξ αρχής να δημοσιευθεί σε αυτή τη μορφή η έκθεση γενικής ανάλυσης. Φυσικά υπάρχουν για κάθε όχημα μια ολόκληρη σειρά στοιχείων του εργαστηρίου που μπορεί να ενδιαφέρουν τους ειδικού που δεν θεωρήσαμε ότι ήταν σκόπιμο να δημοσιευθούν σε αυτή τη φάση. Μπορούμε να δημοσιεύσουμε μια έκθεση πιο λεπτομερή, αλλά σε τι θα εξυπηρετήσει. Υπάρχουν ένα σωρό στοιχεία του εργαστήριου μας. Αλλά δεν αποφασίσαμε να το παρουσιάσουμε έτσι με αυτές τις λεπτομέρειες. Thank you very much. Um, Καταρχήν μια-δυο γρήγορες ερωτήσεις. Πόσοι τύποι αυτοκινήτων ε, ξε, εγκρίνονται αναέτος. Ε, κατά μέσο όρο έχουμε περίπου 300 εγκρίσεις τούπου. Πάνω κάτω. Εντάξει, μπορεί να διαφέρει από χρόνο σε χρόνο, αλλά πάνω κάτω είναι αυτό. Πόσοι από αυτούς τους τύπους είναι οι Ιταλικές μάρκες. E Σχεδόν όλες οι επιστοποιήσεις είναι της Fiat, του ομίλου Fiat. Ναι, έχουμε και άλλες ε, πιστοποίησεις, αλλά ίσως για εμπορικά οχήματα, όμιλος Fiat σημαίνει Fiat, Ferrari, Maserati κτλ. Ε, έχοντας διαβάσει τις γραπτές σας απαντήσεις, αλλά ακούγοντας και αυτό που μας λέτε σήμερα, ως ε, αρχή, ως φορέας. Πιστεύετε ότι εκπροσωπείτε κυρίως, κυρίως λέω, τους πολίτες ή την αυτοκινητοβιομηχανία. Αποστολή μας είναι να εγγυηθούμε την ασφάλεια της κυκλοφορίας των προϊόντων και βεβαίως τον αντίκτυπο στο περιβάλλον. Άρα η απάντησή μου είναι προφανής. Εμείς εργαζόμαστε προς το συμφέρον του πολίτη. Είμαστε μια τεχνική αρχή που καθημερινά ζει Έχουμε επιθεωρήσεις ε, των εγκαταστάσεων, ε, των κατασκευαστών. Η αυτοκινητοβιομηχανία πρέπει να έχει ε, χρόνο προσαρμογής διαφορετικό από αυτό που χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων. είναι πολύ διαφορετικές οι δυναμικές. Χαίρομαι που λέτε ότι δουλεύετε για τα συμφέροντα των πολιτών, αλλά θα σας ρωτήσω, ε, ε τούτου λεχθέντος, είπατε ποτέ όχι σε, μια, σε ένα αίτημα έγκρισης τύπου ε, κριτικάρατε ποτέ την αυτοκινητοβιομηχανία παρκώς ε, στην, στην απάντηση της ερώτησης 5 είπατε ότι θα πρέπει να ε, εξισορροπήσετε την ε, προστασία του περιβάλλοντος ε, με την ανταγωνιστικότητα του τομέα. Ε, οπότε πιο πραγματικά αντιπροσωπεύεται και δεύτερον επικρίνατε επαρκώς, ήσασταν επαρκώς επικριτικός στην αυτοκινητοβιομηχανία, πιστεύετε. Io Εγώ πιστεύω πως έχει βρεθεί η σωστή ισορροπία και απόδειξη γι' αυτό είναι το γεγονός ότι πριν να φτάσουμε στην περίφημη ψήφο της 24ης Οκτωβρίου στην Επιτροπή, εμείς ήρθαμε σε διαβούλευση και με χώρες που συνήθως έχουν τελείως διαφορετική, διαμετρικά αντίθετη θέση με την Ιταλία. Ε, διαπιστώσαμε ότι η κατάσταση που δημιουργεί το, δηλαδή οχήματα τα οποία ε, κυκλοφορούν περισσότερο στους δρόμους, έπρεπε να παρέμβουν. Να παρέμβουμε, λοιπόν, έπρεπε να βρούμε μια συμβιβαστική. Γιατί αν είχαμε υιοθετήσει ένα όριο του ενός, κανένα όχημα δεν θα μπορούσε να πιστοποιηθεί από το 2017. Οπότε, χρειάστηκε να βρούμε κάποια μορφή συμφωνία. Γιατί ακόμα και κάνοντας υπολογισμούς, αποτέλεσμα ήταν ότι οφέλο ε, θα υπήρχε, κέρδος θα υπήρχε Διαφορετικά, θα έπρεπε να μείνει και κάποιο κέρδος, διαφορετικά δεν καταφέρναμε τίποτα. Ε, πριν από δύο εβδομάδες με την EPA ε, συζητήσαμε θέματα συμμόρφωσης και δεν καταλαβαίνουν ε, το τι συζητάμε, διότι αυτοί έχουν ένα επίπεδο ρήπων και αν δεν συμμορφώνεις δεν μπορείς να πάρεις έγκριση τύπου. δεν πιστεύετε ότι υπάρχει τεχνολογία. Όλοι οι εμπειρογνώμονες αυτό λένε. Δεν πιστεύετε ότι θα πρέπει να καταργηθεί η συμμόρφωση και να έχουμε απλώς ένα επίπεδο ρήπων κάτω από το οποίο δεν θα εγκρίνεται κανένα όχημα. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, στη ΣΥΠΑ δεν υπάρχει δοκιμή στο δρόμο. Το να ζητάνε από εμά ε, παράγοντε συμμόρφωση ε, μου φαίνεται πολύ παράξενο. Αν υπήρχε, εντάξει, να το συζητούσαμε, αλλά δεν κάνουν καν ε, δοκιμή στο δρόμο. Ε, πρέπει να το δούμε και πιο θετικά. Εμείς είμαστε πρώτοι στον κόσμο που εισάγουμε δοκιμή στο δρόμο. Οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν. Χώρες όπως η Αυστραλία σε διεθνές επίπεδο μας ζήτησαν να αναπτύξουμε κοινού κανόνες, κάποιο κοινό πρωτόκολλο. Αλλά πολλές χώρες δεν είναι ακόμα έτοιμες γιατί βλέπουν αυτή τη δικασία RDA ως μια πρωτοπόρα ε, διαδικασία για το στόχο πιστοποίησης ε, του αυτοκινήτου, όχι για το αν δουλεύει καλά ή όχι. Τώρα βέβαια με το σκάνδαλο Volkswagen ε, απέκτησε πιο επίγοντα χαρακτήρα. Εγώ θεωρώ λοιπόν πως είναι θετικό αυτό. Ε, κάτι που μας είπε η EPA είναι ότι ε, έχουν διάφορες δοκιμές για να ελέγξουν αυτοκίνητο και πριν την κυκλοφορία του ε, και κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας, και τη διάρκεια δηλαδή της χρήσης του. Ε, μας είπαν επίσης ότι θέλουν να εισαγάγουν και ένα στοιχείο μη προβλεψιμότητας στις ε, δοκιμές έτσι ώστε οι αυτοκινητοβιομηχανίες να μην ξέρουν ακριβώς σε τι δοκιμαστούν. Πιστεύετε ότι είναι μια καλή πρόταση? Δεν κατάλαβα καλά. Ε, είπατε στο test random, στα τυχαία τυχαίες δοκιμές εκτός των κύκλων. Ναι. On the road, ναι. Το, το έχουμε. Αλλά για εμάς τώρα είναι το RDA. Έχουμε μια παράλληλη περίπτωση που ασχολείται με το, με το θόρυβο. Υπάρχει το in-service conformity testing. Το RDA όμως ε, προβλέπεται μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας που χρησιμοποιείται Εκεί μπαίνει και το RDA Δεν είναι μόνο μία αρχή, όπως τις είπα, είναι 28 οι αρχές ελέγχου και πιστοποίησης. Μπορεί δηλαδή ένα ε, όχημα το οποίο ξεπερνά το RDA στην Ιταλία να αμφισβητηθεί από μια άλλη αρχή. Γιατί ίσως να κάνουν εκεί μια δοκιμή, όχι εργαστηρίου, στο δρόμο, ίσως σε διαφορετική διαδρομή μέσα στο πλαίσιο του κύκλου. Αλλά το αποτέλεσμα να διαφέρει και εκεί θα υπάρχουν... Ε, ε, ναι, θα σας διακόψω πάλι. Ε, να σας διακόψω. Ε, έχουμε ένα σύστημα μεταξύ των 28 κρατών μελών για το σύστημα τύπου έγκρισης, έγκρισης αλλά έχουμε και μια καινούργια πρόταση της Κομισιόν και πρέπει να βελτιώσουμε αυτή την πρόταση της Κομισιόν. Ε, υπάρχει και η ιδέα μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας που θα αναλαμβάνει την ε, επιτήρηση της αγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο πιστεύετε ότι είναι μια καλή ιδέα μια τέτοια ευρωπαϊκή υπηρεσία για να κάνει αυτά που δεν κάνουν τα κράτη-μέλη. Εποπτεία τη αγορά θεσπίστηκε ω Γενική Αρχή πριν από κάποια χρόνια. Να σα αφήσω τα κρατη μέλη να το κάνουν. Χρειάζονται πόρου. Εμείς και κάπου πρέπει να τους βρουν. Εμείς το έχουμε κάνει με, μια σωρό, κάποιες που κάνουμε για τα οχήματα, για τα, την ασφάλεια, τα, την των παιδιών, τα κράνη για τις μοτοσυκλέτες κτλ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι ένα πεοχιακό φαινόμενο, αλλά ότι θα σταθεροποιηθεί. Πώ θα το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξέρω. Ε, ε Εμεί έχουμε αμφιβολίε. Θα ήταν καλύτερο τα κράτη-μέλη να συγκεντρώσουν τις αρκετούς πόρους ανθρώπινους και ε, ε, να μπορέσουν να το κάνουν οι ίδιοι. Να μπορούν, δηλαδή, μπορεί να πιστοποιήσει η, η Κομισιόν ότι κάνουν όλοι τον ίδιο έλεγχο. Αλλά τώρα να φτιαχτεί ένα οργανισμό, δεν νομίζω, όχι. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Και από δική μου πλευρά σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήλθατε εδώ πέρα σήμερα να απαντήσετε στις ερωτήσει μα. Θα ήθελα να θέσω το θέμα του παρελθόντο και βάσει των όσων έχω παρακολουθήσει και έχω ακούσει τις τελευταίους μήνες εδώ στην Επιτροπή. Θα ήθελα να ξέρω πώς ε, και για την Ιταλία και για τις άλλε χώρες σε ό,τι αφορά την έγκριση τύπου Συνεργαστήκατε ή δεν συνεργαστήκατε γιατί είναι συγκεκριμένο στοιχείο. Σε ό,τι αφορά δηλαδή οι περιπτώσεις όπου οι κατασκευαστές προσπάθησαν να ξεφύγουν. Για παράδειγμα στην Ιταλία είχαμε τη Fiat. Αλλά θεωρητικά θα μπορούσε να στραφεί και μια άλλη εταιρεία προς εσάς να αποφασίσει μια αυτοκινητοβιομηχανία για παράδειγμα ότι θα πάει στο Λουξεμβούργο ή κάπου αλλού ή εν περιπτώσει όπου είναι πιο ευνοϊκό. Πώς ε, το αποφεύγεται αυτό το φαινόμενο του να πηγαίνει δηλαδή κάθε εταιρεία εκεί που τη βολεύει καλύτερα. Guardi, ε, credo di aver risposto a questa domanda e oh, θα προσπαθήσω να απαντήσω και θα προσθέσω και γραπτό. Στη θεωρία ένας κατασκευαστής δεν μπορεί να υποβάλει δύο ή περισσότερες αιτήσει επιστοποίηση σε διάφορα κράτη. Μπορεί μόνο σε ένα κράτος να το υποβάλει. Όμως, όταν ένας κατασκευαστή έχει αμφιβολίε για μια τεχνική λύση, ας πούμε, στρέφεται σε μια αρχή και ζητά να μπορέσει να πιστοποιήσει αυτού του είδου το όχημα. Αν λάβει αρνητική γνώμη, αποσύρει το αίτημά του και ίσω ναι, μπορεί να στραφεί αλλού για να ζητήσει έγκριση και επιστοποίηση. Αυτό είναι δυνατόν. Εμείς σε ορισμένες περιπτώσεις όπου δώσαμε αρνητική γνώμη, μας είπαν οι συνάδελφοι ότι κάποιες φορές πήραν την έγκριση από άλλες αρχές. Θα ε, πρέπει να πω ότι εμείς, αλλά όχι γιατί είμαστε κρατική, κρατικός οργανισμός, δηλαδή δεν έχουμε κέρδος το κέρδος μάλλον ως βασικό μας στόχο, οπότε συχνά δεν δίνεται η πιστοποίηση. Και φεύγουν. Τώρα αν στραφούν σε άλλη χώρα, αυτό δεν το ξέρουμε σε πάντα. Κάποιες φορές μας ενημερώνουν. Συγγνώμη, είναι σημαντικό το εξής. Συνήθω εμείς συνομιλούμε με τις άλλε αρχές. Όταν ένας κατασκευαστή μας προβάλλει μια λύση, εμείς στέλνουμε mail στις άλλε αρχές και ρωτάμε, λέμε, ορίστε, αφού μας προτείνουν αυτή τη συντεχνική λύση. Για κατά τη γνώμη σα αυτό είναι δυνατόν ή όχι. Εμείς το βρίσκουμε δύσκολο. Εσείς τι λέτε. Σας ευχαριστώ. Μία σύντομη δεύτερη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, σε ό,τι αφορά τι δειγματοληπτικές ε, δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ό,τι αφορά τα οχήματα που έχουν ήδη λάβει έγκριση τύπου. Έχει αλλάξει τίποτε από το που ξέσπασε το σκάνδαλο. Κάντε μήπω πιο πολλέ ε, τέτοιε δοκιμέ και πιο πολλού τέτοιου δειγματοληπτικού ελέγχου από το που ξέσπασε το σκάνδαλο. Έχει αλλάξει κάτι. Tanto δοκιμές που κάναμε στην Νάπολη και στο Τωρίνο, που είναι ένα στοιχείο για να δούμε πώς ε, συμπεριφέρονται τα οχήματα Euro 5. Τώρα, Γίνονται οι δοκιμές για την ασφάλεια και τις εκπομπές και συνεχίζουμε να κάνουμε τους ελέγχους συμμόρφωσης του προϊόντος. Πρόκειται για την παραγωγική διαδικασία, την ποιότητα μάλλον της ε, παραγωγικής διαδικασίας, πάμε και ελέγχουμε διάφορες ε, εγκαταστάσεις κατασκευαστών για όλα τα στοιχεία. Ο κ. Γερμπράντη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, στην Επιτροπή αυτή ε, έχουμε ενδείξεις ότι κάποια πολλά κράτη-μέλη ε, έχουν επιφυλάξεις στο να εργαστούν υπέρ του περιβάλλοντος ενώπιον της δικής του Μία από, αυτή, μία από αυτές τις χώρες είναι η Ιταλία. Ε, η Fiat για παράδειγμα ε, είναι μέλος σε πολλές ε, τεχνικές επιτροπές. Η Ιταλία πολύ συχνά προσπαθεί να επιβραδύνει διαδικασίες αντί και LTP οι Ιταλικές ε, αρχές ε, παρεμβαίνουν ιδιωτικώς ενώπιον της Fiat και δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ε, το ερώτημά μου είναι γιατί επιτρέπεται στην Fiat να σβήνει εν μέρη το σύστημα κυκλοφορίας καυσαερίων. Σύμφωνα με την Ιταλική μελέτη τα ε, αυτοκίνητα της Fiat δεν εκπέμπουν 20 φορές περισσότερο, περισσότερο οξύδια του αζότου, αλλά, όπως στη Γερμανία, αλλά 6, 6 φορές περισσότερο από το όριο. Αυτό σημαίνει ότι εσείς θα έπρεπε να αναλάβετε αμέσως δράση. Είπατε στη Fiat ποτέ ότι θα αποσύρετε την έγκριση τύπου αν δεν διορθωθεί αυτό σε ένα σύντομο ε, και το χρονικό διάστημα. Τι κάνατε για να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Εμείς δεν μπορούμε να αποφέρουμε καμιά πιστοποίηση γιατί, επαναλαμβάνω, ο έλεγχος πιστοποίησης από εμά είναι θετικός. Εμείς ε, πιστοποιούμε επί τη βάση συγκεκριμένου πρωτοκόλου. Εμείς γνωρίζουμε τα όσα συμβαίνουν εκτός του κύκλου του ελέγχου. Συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά σύμφωνα με τη Γαλλική και την Ολλανδική Αρχή Πιστοποίησης πρόκειται για ένα σαφές παράδειγμα μιας παράνομης συσκευής αναστολής. Μπορείτε ευκολότατα να ρωτήσετε τι ΦΙΕ τι κάνει και γιατί και μετά να κρίνετε αν είναι παράνομο ή όχι. Ή μπορεί να ρωτήσετε από τους Γάλλους και τους Ολλανδούς συναδέλφους γιατί πιστεύουν ότι πρόκειται για μια παράνομη συσκευή αναστολής. Πρώτα απ' όλα, δεν συναντήσαμε καμία τέτοια συσχεδία. Έχουμε στείλει την έκθεση μας στην KBA. Ε, αυτή δεν συμφωνεί, εντάξει. Μα εντυπωσίασε ε, η στάση τη. Αντί να μα στείλει ε, επιστολή και να μα πει δεν συμφωνούμε μαζί σα, έστειλε επιστολή στην Κομισιόν και λέει η Ιταλία κάνει διαφορετική, μάλλον έχει διαφορετική γνώμη και η Κομισιόν βρίσκεται να κάνει το διαιτητή υπό φυσιολογικέ συνθήκες εμεί περιμέναμε μία απάντηση τέτοιου τύπου. Ε, δεν συμφωνούμε, ας τα πούμε από κοντά στη Ρώμη ας πούμε ή στο Βερολίνο. Τώρα, για τους γαλλικέ αρχές δεν λάβαμε ποτέ γραπτή ανακοίνωση από πλευρά των γαλλικών ή των γερμανικών αρχών που να μας λένε ότι για μας αυτά τα οχήματα δεν είναι νόμιμα. Το έκανε μόνο η KBA μέσω τη Κομισιόν, θα το συζητήσουμε το Νοέμβριο με την Κομισιόν. Mm, εσείς όμως τι κάνατε με τη Fiat, ο, είδατε ότι αυτό το 500 XL, το Fiatάκι το 500 XL εκπέμπει τόσες πολλές ρήπους. Συζητήσατε με τη Fiat, τους είπατε να λύσουν το πρόβλημα. Δεν το κάναμε από την νομική άποψη, γιατί δεν μπορούμε να ζητήσουμε από έναν κατασκευαστή οχήματος να παρέμβει, γιατί την έχει την πιστοποίησή του. Την... να αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οποιαδήποτε παράνομη συσκευή αναστολή η οποία δεν ε, εντοπίζεται σε EDC δεν μπορεί να εντοπιστεί από τι ταλικέ Αρχέ. Και ακόμα, ακόμα μα λέτε ότι είναι και παράνομο ακόμα να την ε, ανακαλύψει κανείς έτσι. Είναι περίεργο, περίεργο, περίεργο αυτό και νομίζω ότι επιβεβαιώνει το παράδειγμα που σας το πρωί. Ναι, όχι, όχι, όχι, δεν έχει τίποτα το παράξενο. Στην υπόθεση τη Fiat και δεδομένων των διαμαρτυριών τη ε, της Γερμανίας κάναμε και δοκιμέ εκτός του κύκλου ε, με διαφορετικέ θερμοκρασίε και στο δρόμο. Εκτό κύκλου το ελέγξαμε το διαπιστώσαμε ότι αυτό το όχημα εκπέμπει περισσότερο επειδή συμπεριφέρεται ομοιόμορφα τόσο στο δρόμο όσο και στο εργαστήριο. Συμπέρασμα μα είναι ότι δεν υπάρχει defeat device. Γιατί αν υπάρχει defeat device αλλάζει η συμπεριφορά. Εδώ δεν αλλάζει τίποτα. Εκπέμπει το ίδιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό... Μα είναι αδύνατον γιατί το τεστ είναι 20 λεπτά μόνο στα 22 λεπτά τι σε 22 δεν εμφανίζεται σε ένδυση. Άρα πώς έχει την ίδια συμπεριφορά στις δοκιμές και στον δρόμο το όχημα lo sappiamo bene, ma eh, se la norma oggi Το γνωρίζουμε καλά, αλλά ο κανόνα τι μα λέει. Μα λέει να ελέγξουμε ένα οχήμα ε, στο εργαστήριο. Αλλά θα πρέπει να είναι αυτό σύμμορφο και προ τι φυσιολογικέ συνθήκε χρήση, οι οποίε ορίστηκαν τώρα μόνο με το RDE. Τότε δεν μπορούσαμε εμεί να παρεύουμε. Ναι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η κατάσταση. Το λέει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υιοθέτηση της διαδικασίας ΣΕΡΔΙΕ. Αυτή είναι η δοκιμή για να επαληθεύσουμε αν ένα όχημα είναι φυσιολογικό στις φυσιολογικές συνθήκες χρήσης. Διαφορετικά πρέπει ένα όχημα να το ελέγξουμε υπό κάθε δυνατή συνθήκη. Ε, στο βουνό, στο λόγκο, στο βόρειο πόλο και... Τι να κάνουμε άλλο. Ευχαριστώ. Σάλβα. Ε, Ευχαριστώ. Θα επανέλθω στην πρώτη μου ερώτηση. Ε, δεν Είπατε ότι δεν υπήρχαν ε, μεταξύ των διαφόρων χωρών διαφόρες στην εφαρμογή των κανόνων συμμόρφωσης. Οπότε πώς εξηγείτε ότι μια χώρα όπως το Λουξεμβούργο που δεν έχει αυτοκινητοβιομηχανία δική του λαμβάνει τόσες αιτήσει, τόσα αιτήματα έγκρισης τύπου. Οι αρχές ε, του Λουξεμβούργου ε, θα μπορούν να το εξηγήσουν. Εμείς από τον έλεγχο γνωρίζουμε ότι το Λουξεμβούργο έχει διάφορες, ε, έχει έρθει σε επαφή με διάφορες τεχνικές ε, υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Λειτουργούν για το Λουξεμβούργο. Ε, και υπάρχει μία λυσίδα ε, επιχείρησιακή τουρκική ανάμεσα στι χώρε. Τώρα, αν ε, στο συγκεκριμένο εργαστήριο του Λουξεμβούργου κατήσατε υπεύθυνο ενώπιον όλων των άλλων αρχών για την λειτουργία υπάρχει μια αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ μας. Το Λουξεμβούργο μπορεί να οργανωθεί με τον τρόπο που θεωρεί σωστό σεβόμενο πάντοτε τους κανόνες της οδηγίας πλαισίου που είναι πολύ συγκεκριμένους όσον αφορά τα, στάνταρ που πρέπει, τα ποιοτικά στάνταρ που πρέπει να γίνονται σεβαστά. Ναι, αλλά είναι πολύ πιθανό το Λουξεμβούργο να χρησιμοποιεί άλλες υπηρεσίες που δεν είναι στην επικράτειά του. Ε, άλλη ερώτηση και επιστρέφω στη δεύτερη ερώτηση που σας είχα κάνει στην αρχή σε ό,τι αφορά τις νέες διαδικασίες έγκρισης τύπου. Ε, ποια είναι η δική σας αξιολόγηση, θα προσαρμοστεί εύκολα η αυτοκινητοβιομηχανία. Γιατί ε, προηγουμένως εκφράσατε κάποιες αμφιβολίες. Ε, είχατε πει ότι είναι μια διαδικασία από τεχνική πλευρά πολύ περίπλοκη. Θα είναι εύκολο η αυτοκινητοβιομηχανία να προσαρμοστεί γρήγορα και ποιες συνέπειες μπορεί να έχει στο κομμάτι των κινητήρων diesel, ε, ιδιαίτερα στην Ευρώπη που η οποία πρώτο στατεί, είναι πρωτοπόρος σε θέματα κινητήρων diesel στην αυτοκίνητα βιομηχανία. Ξεκινάμε από την προϋπόθεση ότι η ε, ευρωπαϊκή βιομηχανία για ένα σωρό είναι υποχρεωμένη να παράγει ποιοτικά αυτοκίνητα diesel για παραγωγές ε, μεγάλης ε, κλίμακας. Αναμένοντας ε, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το diesel παραμένει η λύση για την ώρα. Γι' αυτό οι κατασκευαστές πρέπει να καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες, ιδιαίτερα αυτοί που κατασκευάζουν πιο μικρά αυτοκίνητα, για να μπορέσουν μέσα σε μικρά αυτοκίνητα και λιγότερο δαπανηρά αυτοκίνητα να εντάξουν ένα σωρό μηχανισμούς, ώστε το αυτοκίνητο να σέβεται τα όρια εκπομπών σε κάθε συνθήκη οδήγησης. Δηλαδή πιο εξελιγμένες τεχνολογίες, αυτή που λέγεται SCR. Ε, είναι τεχνολογίες ε, που ε, θα πρέπει να προσαρμοστούν και στα μικρότερα αυτοκίνητα. Μπορεί, ας πούμε, ένας κατασκευαστής να μην φτιάχνει διζελοκινητήρες για τα μικρά αυτοκίνητα, αλλά να φτιάχνει, ας πούμε, κινητήρες με αέριο. Το έχουμε διαπιστώσει και σε κατασκευαστές μη Ιταλούς αυτό. Ευχαριστώ, κυρία Ντέλη. Κύριε Ρέριο, σας ακούω εδώ και ώρα. Θέλω να σχολιάσω διάφορα. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την απάντηση στην ερώτηση 9. Λέτε δεν υφίσταται ορισμός κανονικής χρήση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι εκπομπέ. Ε, ισχύει αυτό και για τα φρένα. Τι πιστεύετε. Ποια είναι η όψη σα. Μιλώ για τα φρένα των οχημάτων. Βλέπετε ότι υπάρχει ορισμός για την κανονική χρήση ή όχι. Ναι, βεβαίω. Αλλά η δοκιμή για το φρενάρισμα γίνεται πάντα σε αληθινές συνθήκες οδήγησης. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο φρένα και στις εκπομπές του οχήματο. Η συμπεριφορά ενός οχήματο σε πίστα είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα, γιατί για τα φρένα λοιπόν είναι σωστό όπως γίνεται, διαφορετικό είναι για τις εκπομπές και συγγνώμη αν το επαναλαμβάνω, αλλά η δοκιμή RDE είναι ε, πολύ σημαντική γιατί κανένας άλλος δεν τη κάνει. Ευχαριστούμε και το Κοινοβούλιο που το έκανε γιατί αν δεν το είχε κάνει ακόμα θα συζητούσαμε. Λέτε κύριε Ράριο ότι είναι δυνατόν να γίνουν δοκιμές οδήγησης στο δρόμο για τα φρένα αλλά όχι για τα καυσαέρια και τις εκπομπέ. Τέλο πάντων, το αφήνω αυτό. Κατά την άποψή σα. αν κατάλαβα καλά, η δική σα αποστολή είναι να εφαρμόζετε τι ε, δοκιμέ του κύκλου για τη συμμόρφωση, ε, αλλά όχι ε, τη συμμόρφωση με όρια σε οικονομικέ συνθήκες. 75.000 ε, ε, άτομα το χρόνο πεθαίνουν όμως από εξαιτία υψηλών, ορίων, υψηλών εκπομπών οξυδίων του αζότου. αν γινόντουσαν όμως σεβαστοί οι κανόνες πολλοί θα είχαν γλιτώσει τη ζωή τους. 21.000 από αυτούς τους ανθρώπους είναι Ιταλοί. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η αποστολή σας είναι να εφαρμόζετε και να εξασφαλίσετε ότι θα ε, γίνονται σεβαστοί οι κανόνες στο σύνολό τους και όχι μόνο οι ελάχιστοι κανόνες για την πιστοποίηση και την έγκριση τύπου. Δεύτερον, τι κάνατε για να εγγυηθείτε την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα οχήματα συμμορφώνονται με τα ανώτατα όρια. Ευχαριστώ. Ίσως να μην εξηγήθηκα καλά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Σήμερα οι δοκιμές για τις εκπομπές γίνονται σε εργαστήριο. Μεθαύριο το 2017 θα γίνεται με το RDE στο δρόμο για το φρενάρισμα ε, ανέκαθεν. Ναι, οι δοκιμές γίνονται στο δρόμο. Το RDA μόλις τώρα φτιάχτηκε το 2017. Παλιότερα οι δοκιμές γίνονταν αποκλειστικά στο εργαστήριο και είχαν απλά συγκριτικό χαρακτήρα. Γιατί δεν εφαρμόσαμε το άρθρο 5. Εμείς το άρθρο 5 προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα που επαναλαμβάνω από την άποψη της εφαρμογής και αναφέρομαι στους κανονισμούς της Κομισιόν δεν έχει καμιά αναφορά. Αυτό δεν σημαίνει δηλαδή, δηλαδή δεν υπήρχε καν υποχρέωση για τον κατασκευαστή να δηλώσει ποια στρατηγική εκπομπών ε, υιοθετούσε. Αυτή η υποχρέωση προκύπτει μόνο με το RDE. Το σύστημα για τα βαριά οχήματα δεν υπήρχε για τα αυτοκίνητα, τα γιοταχή. Περισσότερο τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ρωτηθούν. Τώρα έχουμε ευθυγραμμιστεί και με το RDE πρέπει οι κατασκευαστές να δηλώνουν τη στρατηγική. Παλιότερα δεν ήταν αυτό υποχρεωτικό. Mr. Erario. Κύριε Ράριο, τελειώνουμε αυτήν την ακρόαση, ε, αλλά υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι η ΕΦΙΑ θα είναι μαζί μας εδώ την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε πολλές από τις ερωτήσεις που ε, δεν απαντήθηκαν σήμερα μπορούν να απαντηθούν την επόμενη εβδομάδα. Ε, Έχουμε και γραπτή διαδικασία για πρόσθετες ερωτήσεις. Ε, κάθε απάντηση εγείρει καινούργια ερωτήματα. Ε, μέχρι τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου παρακαλώ πολύ που βάλει τις ερωτήσεις σας στον κύριο Εράριο. Ευχαριστούμε κύριε Εράριο. Ε, ευχαριστούμε που προσπαθήσατε να απαντήσετε σε δύσκολες ερωτήσεις. Και ο κύριος Εράριο ευχαριστεί. to keep track of our timing. Ε, για να μην ε, χάσουμε ε, την παρακολούθηση του χρόνου θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Άλεξ Μπέρνς να καλωσορίσω τον κύριο Άλεξ Μπέρνς εκτελεστικό διευθυντή της Millbrook Group έχει ήδη ζεσταθεί παρακολουθώντας το πρώτο τμήμα της, την πρώτη ακρόαση παρακαλώ πολύ έχετε το λόγο για 10 λεπτά δεν θα μου πάρει παραπάνω από δύο λεπτά εισαγωγή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Παρακαλώ πολύ συνάδελφοι, ησυχία. Ε, Εκπροσωπώ την Μιλμπρουκ, το, τον όμιλο Μίλμπρουκ, είναι ένας πάροχος υπηρεσιών δοκιμών ε, προς την αυτοκινητοβιομηχανία. Ε, έχουμε γραφεία στον Ηνωμένο Βασίλειο και τη Φιλανδία, είμαστε ανεξάρτητοι, αμερόληπτοι ε, και τα, οι δοκιμές μας υποβάλλονται σε εξωτερικούς ελέγχους. Ε, εργαζόμαστε από το 1970 και συγκρίνουμε τα αποτελέσματά μας με αυτά άλλων παρόχων προκειμένου να ε, είμαστε σίγουροι για την αποτελεσματικότητά μας. Ε, δίνουμε, προπαρέχουμε αποτελέσματα δοκιμών στην ανάπτυξη οχημάτων και στην πιστοποίηση. Ε, η πιστοποίηση οχημάτων είναι ένα μικρό κομμάτι του συνολικής μας ε, δουλειάς. Παρέχουμε επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες περιορισμένες ε, που βοηθάει, βοηθούν μικρές εταιρείες να καταλάβουν τις δοκιμές μας όχι, δεν δίνουμε όμω συμβουλευτικέ για το πώ θα περάσουν αυτέ τι δοκιμέ οι εταιρείε αυτέ. Επίση, βοηθάμε στην ανάπτυξη κύκλων δοκιμών που να αντιπροσωπεύουν πραγματικέ συνθήκε οδήγηση και χρησιμοποιούνται συνήθω για την ανάπτυξη λιγότερο ρηπενών των οχημάτων ρηπογόνων οχημάτων. Για παράδειγμα, ε, τον ε, ε, Millbrook London Bus, Transport Bus Cycle, που είναι κύκλος δοκιμών για λεωφορεία που χρησιμοποιούνται από τη μεταφορική εταιρεία του Λονδίνου. Ε, για δοκιμές πιστοποίησης η Milbrook συνήθως ε, λειτουργεί ως εργαστήριο ε, ενώ η VCA του Ηνωμένου Βασιλείου Vehicle Certification Agency δρά ως τεχνική υπηρεσία και φορέας έγκρισης τύπου. Αυτό σημαίνει ότι η ακυρότητα των δοκιμών μας ελέγχεται από την VCA. Ε, το, ε, η λειτουργία των δοκιμών, η ενέργεια των δοκιμών ορίζεται από κανονισμούς και ως εργαστήριο εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την ε, ε, για να γίνονται οι δοκιμές ε, και τα αποτελέσματα είναι αξιόπιστα, όχι όμως για να αποφασίζουμε αν η α ή β δοκιμή είναι κατάλληλη ή όχι. Ε, μάλιστα το μοντέλο, το μοντέλο βασίζεται στην ανεξαρτησία μας και οποιαδήποτε υποψία, υπόνοια ε, ότι αυτή δεν λειτουργεί σωστά θα αποτελούσε σημαντική σκιά στη λειτουργία μας και στο όλο τομέα. And, uh, Ευχαριστώ κύριε Μπέρντς για τις παρατηρήσεις σας. Πριν από δύο-τρεις εβδομάδες ε, ε, επισκέφθηκαν την Επιτροπή μας κάποιοι συναδελφοί μας από το Λουξεμβούργο και τη Γερμανία. Μάλλον ορισμένοι μας συναδελφοί επισκέφθηκαν το Λουξεμβούργο και τη Γερμανία ε, και αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο τον κόσμο των, των εγκρίσεων τύπου και των τεχνικών δοκιμών. Ένας από τους ε, μία πραγματικότητα είναι, που με ενοχλεί μάλιστα είναι ότι η όλη διαδικασία συμμόρφωσης ε, Ε, είναι η διαδικασία συμμόρφωσης. Εσείς ε, ε, έχετε τέτοιου είδου δραστηριότητες. Ναι, ορισμένες από τις δοκιμές που κάνουμε για κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν σχέση με συμμόρφωση διαδικασιών παραγωγής. Ε, επόμενη ερώτηση. Ε, και ε, είστε ενεργοί και σε θέματα παρακολούθηση αγοράς. ναι, μπορούμε να το κάνουμε, αλλά δεν μας έχει ποτέ ανατεθεί. Εδώ και κάποια χρόνια τουλάχιστον μας έχει ανατεθεί. Σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση παραγωγής, αν κατάλαβα καλά, ε, Ε, γίνονται η δουλειά, η περισσότερη δουλειά γίνεται από τους ίδιους τους, από τους ίδιους κατασκευαστές, δεν είναι και ελέγχεται μετά. Ε, ένα στοιχείο δεν ελέγχεται καθόλου και αυτό είναι το λογισμικό, είναι αλήθεια. Χωρίς μικρόφωνο μιλτής. Ο, αυτοκίνητο, ε, ο κατασκευαστής μας παρουσιάζει ένα αυτοκίνητο το οποίο εμείς δοκιμάζουμε το αυτοκίνητο έτσι όπως μας παρουσιάζεται. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται δοκιμή του λογισμικού. Εννοώ ότι ε, όταν ένα αυτοκίνητο μπει στην παραγωγή και ο κατασκευαστής χρειάζεται να πάρει την έγκριση μόρφωσης ε, περνούν κάποιοι μήνες ανάμεσα στην, ε, πρώτη ε, έγκριση τύπου και την ε, εμπορία, θέση σε εμπορία του αυτοκινήτου. Εν τω μεταξύ, το λογισμικό ενδεχομένως μπορεί να αλλάξει και τελείως. Και στην ενδιάμεση αυτή περίοδο δεν γίνεται έλεγχος του λογισμικού. Με την ε, δήλωση συμμόρφωσης ε, παραγωγής ε, δεν γίνεται έλεγχος για το κατά πόσο το λογισμικό λειτουργεί σωστά όπως λειτουργούσε τη στιγμή που δόθηκε η, έγκριση, η ερκή έγκριση. Αυτό μπορεί να ισχύσει και για το hardware. Δηλαδή ο κατασκευαστής θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το αυτοκίνητο το οποίο εμπορεύεται τελικά είναι ίδιο ακριβώς με αυτό το για το οποίο ελήφθη η έγκριση τύπου. Αν δεν είναι θα πρέπει να επανυποβληθεί έτοιμα έγκριση τύπου. Ερώτηση. Με τη δική σας γνώση και επίρα. Πιστεύετε ότι ε, Δίνοντα τέτοιου είδου ευθύνε και ενδεχομένω και νομικέ ευθύνε στου κατασκευαστές ε, είναι σωστό το να δίνουμε τέτοιου ευθύνε, είναι σωστό ε, δεν κατάλαβα να σα ξανακάνω μια ερώτηση ο ρόλος των κατασκευαστών είναι τεράστιος σε αυτή τη διαδικασία πιστεύετε ότι είναι υπερβολικά μεγάλος θα μας συστήνατε να αλλάξουμε αυτή τη διαδικασία στο μέλλον να, να τη βελτιώσουμε απάντηση ε, οι κατασκευαστές από όσο γνωρίζω δουλεύουν σκληρά προκειμένου να συμμορφώνονται με τους ε, κανονισμούς και την ομοθεσία. Η δουλειά τους είναι δύσκολη και γενικά είναι επιμελής σε αυτή τους την προσπάθεια. Δεν έχουμε διαπιστώσει ε, περιπτώσεις ή υπόνοιες ή ενδείξεις ε, υπερβάσεων. Ε, επόμενη ερώτηση. Ε, διαφορές ανάμεσα στις ε, εργαστηριακές δοκιμές και στις πραγματικές εκπομπές. φαντάζομαι το γνωρίζετε αυτό τα τελευταία δύο χρόνια. Ναι, περισσότερο από τα δύο χρόνια. έχετε αντιδράσει ενημερώνοντας τις αρχές, για παράδειγμα, ή κάτι άλλο, προκειμένου να εντοπιστεί αυτή η αυξανόμενη διαφορά μεταξύ των δύο. ναι, το εντοπίσαμε και μας ζητήθηκε να κάνουμε δοκιμές για να επιβεβαιωθούν ε, οι μελέτες που είχαν δημοσιευθεί. Ε, πράγματι εντοπίσαμε αλλαγή και διαφορές και ανάμεσα στον, στα αποτελέσματα του κύκλου NDC και, άλλους, και άλλων κύκλων. Ε, η ανάπτυξη των αυτοκινήτων και η χρήση των αυτοκινήτων έχουν αλλάξει. Ε, δηλαδή έχει αλλάξει πάρα πολύ και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους ε, οι ε, χρήστες. Οπότε ίσως το NEDC να έχει Ε, Ευχαριστώ και ο Σάλβα. Ε, κοιτώντας προς τα πίσω, να ρωτήσω το εξής. Αν η ευρωπαϊκή νομοθεσία ήταν πιο αυστηρή. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο λέω. Τι θα είχε γίνει. Θα είχε συμβεί αυτό που, έχει, που βλέπουμε να έχει συμβεί τώρα. Αν είχαμε ορίσει στο παρελθόν ε, και άλλους κύκλους πιο σύγχρονους, τότε τα αυτοκίνητα θα είχαν συμμορφωθεί. Κάθε φορά που ορίζουμε καινούριου κανόνες, περιμένουμε από την αυτοκινητοβιομηχανία να προσαρμοστεί. Και αν οι κανονισμοί από την άλλη μεριά ε, υπολείπονται των εξελίξεων στην αυτοκινητοβιομηχανία, αναπόδραστα δημιουργείται ένα κενό ανάμεσα στα εργαστηριακά αποτελέσματα δοκιμών και στην πραγματικότητα. Ερώτηση. Πότε υποπτευθήκατε τη χρήση τέτοιων ε, διατάξεων ε, ε, αναστολής όταν το ακούσατε, το διαβάσατε στον τύπο ή νωρίτερα ε, είχαμε μας εξέπληξε το σκάνδαλο μας εξέπληξε πραγματικά ξέραμε ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα τις αριστειακές δοκιμές και την πραγματικότητα. Ε, αλλά αυτή την διαφορά την αποδίδαμε σε έξυπνες κινήσεις των κατασκευαστών, έξυπνες επιλογές των κατασκευαστών, νόμιμες όμως, προκειμένου ε, να κάνουν τα αυτοκίνητά τους τεχνολογικά πιο προηγμένα. Ερώτηση. Πιστεύετε ότι η απαντήσεις της Κομισιόν ε, είναι αρκετές για να αποφύγουμε την επανάληψη τέτοιων σκανδάλων. Είναι δηλαδή επαρκώς φιλόδοξες οι προτάσεις Κομισιόν για να αποφύγουμε την επανάληψη. Πιστεύω ότι η υιοθέτηση των, ε, του κύκλου WLTP, του Παγκόσμιου ε, ε, εναρμονισμένου κύκλου και οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες ε, θα είναι αρκετές. Ε, Παρ' όλα αυτά, οι κανονιστικές αρχές θα πρέπει να παραμείνουν σε γρήγορση διότι οι διαδικασίες θα πρέπει να εξελίσσονται όπως ακριβώς εξελίσσεται και η παραγωγή των οχημάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκλίκε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την κυρία Μπέρνση που μας αφιερώνει τον χρόνο αυτό σήμερα και σας ευχαριστούμε και για τις γραπτές σας απαντήσεις στις ερωτήσεις μας. Να αναφερθώ στην εισαγωγική ερώτηση των δύο εισηγητών. Το θέμα του λογισμικού διευκρινίστηκε. Αυτή η Επιτροπή συστήθηκε σε ό,τι αφορά τις ε, ατασταλίες στη χρήση του software, του λογισμικού. Αλλά είπατε ότι σε ό,τι αφορά το λογισμικό θεωρείται ότι εμπίπτει στην ε, αρμοδιότητα και στην ευθύνη του κατασκευαστή. Και ότι θα πρέπει να ακολουθεί φυσικά νομοθεσία. Αλλά για την περαιτέρω νομοθεσία και τι περαιτέρω διαγραφέ είναι σημαντικό όχι μόνο να υπάρχει εμπιστοσύνη, αλλά να υπάρχει και δυνατότητα ελέγχου εσεί ω ανεξάρτητο εργαστήριο ελέγχου μπορείτε να απαιτήσετε πιο πολύ διαφάνεια σε ό,τι Θα μπορούσατε με επαρκείς ε, εμπειρογνώμονες όχι μόνο να δημιουργήσετε συνθήκες εμπιστοσύνης, αλλά να ελέγχετε και παραπάνω. Ευχαριστώ. Είναι περίπλοκο το θέμα αυτό, γιατί νομίζω ότι οι δοκιμές ε, με διαφορετικά και βάσεις. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε, δεν μας το ζητάει άλλωστε και η νομοθεσία για τους ελέγχους. Δεν έχουμε λοιπόν τέτοια ικανότητα. Θα μπορούσαμε να την αποκτήσουμε, θα μπορούσαμε ενδεχομένω, δεν ξέρω να σας πω, δεν είμαι και ειδικό για τα θέματα αυτά. Αλλά αν δεν υπάρχει ε, τέτοια νομική προδιαγραφή για να γίνονται αυτές οι επιθεωρήσεις για το CLP, θα μπορούσαμε να βρούμε μια τεχνική λύση για την ε, διενέργηση των ελέγχων, αλλά αυτό θα πρέπει να το προδιαγράψουν σε πρώτη φάση και τα νομοθετικά κείμενα. Ερώτηση. Δηλαδή, θα ήσασταν θερτικά σε θέση σήμερα να διενεργήσετε ένα τέτοιο έλεγχο λογισμικού ή όχι. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν περιμένετε να αλλάξει η νομοθεσία, αλλά θα χρειάζεστε και του απαραίτητου πόρου φαντάζομαι. Δεν του έχετε στη διάθεσή σα. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά ακριβέ. Θα έπρεπε να υπάρχει μια επαρκή χρονική περίοδο για οργανώσει όπω η δική μα να αναπτύξουν το δυναμικό αυτό, να αναπτύξουν την ικανότητα αυτή για την διενέργεια τέτοιων ελέγχων. Μάλιστα, ερώτηση πάλι. Σε ό,τι αφορά το θέμα λογισμικό, καλυφθήκαν. Σε ό,τι αφορά το hardware τώρα, το υλικό, λέτε στην απάντησή σας υπαριθμών 4 ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες ε, ενδεχομένως να προωθήσουν κάποιες εγκρίσεις τύπου επειδή υπάρχει διαφορετική εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Αυτό το διευκρινίζεται και προηγουμένως στην ε, ακρόαση του Ιταλού συναδέλφου σας διαπιστώσαμε ότι υπάρχει όντως διαφορετική εφαρμογή της κοινωτικής νομοθεσίας και μόνο μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας να κοιτάξουμε δεν είναι ίδια η εφαρμογή του κινητικού δικαίου. Εσείς έχετε κάποια διαφορετικά παραδείγματα για την διαφορετική αυτή εφαρμογή του κινητικού δικαίου. Απάντηση. Καταρχάς να κοιτάξουμε τι, πόσα τεστ, πόσοι έλεγχοι χρειάζονται για να περάσει και να πάρει ένα όχημα έγκριση τύπου από τις αρχές. Η συνάντηση ενδεχομένω μεταξύ του βιομηχανού και τη εταιρεία δηλαδή και τη υπηρεσία ε, έγκριση, χορήγηση έγκριση και πόσοι έλεγχοι χρειάζονται προτού το όχημα όντω πάρει έγκριση τύπου. Όλα αυτά λοιπόν θα συζητηθούν και εδώ πραγματικά μπορούμε να δούμε διαφορετικές εφαρμογές από τις διάφορες υπηρεσίες έγκρισης τύπους. Τα αποτελέσματα όμως του ελέγχου δεν ε, ερμηνεύονται με διαφορετικό τρόπο. Γιατί είναι σαφή, σαφής οι διπροτεγραφές. Γίνεται ο έλεγχος, καταγράφονται τα αποτελέσματα και κατατίθενται. Ευχαριστώ κυρία Νταλή. Σας ευχαριστώ πρόεδρε Κανένα πρόβλημα. Απαντάω και στα δύο ονόματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μπέντε, που είστε εδώ μαζί μα σήμερα στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ και για τις πληροφορίε που μας δίνετε. Να εστιαστώ στην απάντηση στι υπαριθμών 6. Αναφέρεται ότι τα οχήματα ακολουθούν τις τεχνικές προδιαγραφές ε, του κατασκευαστή και όπως ορίζουν και οι υπηρεσίες τις σχετικές. Θα μπορούσα ότι σας παρακαλώ να μας δώσετε πιο πολλές πληροφορίες. Οι κατασκευαστές έχουν την ευελιξία για να προσαρμόσουν τα οχήματά τους σε ό,τι αφορά την έγκριση τύπου, γιατί είναι λίγο ανοιχτό και κρεμές αυτό το ερώτημα. Απάντηση. Υπάρχουν πολύ περιορισμένοι τομείς στους οποίους ε, το όχημα μπορεί να μεταβληθεί για την έγκριση τύπου. Ένα από αυτά είναι και η πίεση των ελαστικών. Γιατί οι συσκευές ελέγχου στο εργαστήριο είναι σημαντικό για να λειτουργήσουν να υπάρχει σωστή πίεση, υψηλή πίεση των ελαστικών. Σε κάποιου τέτοιου τομεί, λοιπόν, ενδεχομένω να υπάρξει κάποια τροποποίηση του οχήματο προκειμένου να α, μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκε της, ε, του ελέγχου στο εργαστήριο, γιατί είναι διαφορετικές οι συνθήκες αυτές από ότι οι συνθήκες ε, στο δρόμο. Αναφέρθηκε από εμπειρογνώμονα ερώτηση ότι ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες ε, απώλειες στις δοκιμές στο εργαστήριο. Το γεγονός λοιπόν ότι υπάρχει αυτό το περιθώριο α, ελιγμού ανταποκρίνεται τελικά, αποτυπώνει τις συνθήκες που επικρατούν στον δρόμο. απάντησε, Χρειάζεται ένα σύστημα ασφαλούς ελέγχου των οχημάτων. Αν δεν υπάρχουν μέθοδοι, αν δεν υπάρχουν λόγοι ειδικοί για τους οποίους πρέπει να τροποποιηθεί ένα όχημα για να μπορεί να ελεγχθεί και αν αυτό περιορίζει τις εκπομπές, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά. Αναφέρεται όμω ε, στην πίεση των ελαστικών. Τι άλλα περιθώρια λιγμού έχει ο κατασκευαστή σε ό,τι αφορά τι τεχνικέ προγραφέ αυτέ. Πολύ περιθώριο, πολύ περιορισμένο περιθώριο. Όπω, δεν είμαι εμπειρογνώμονα, δεν είμαι ειδικό σε τέτοια θέματα. Ε, Ενδεχομένω να υπάρχουν θέματα για το πόσο φορτισμένη είναι η μπαταρία κτλ. Αυτά όμω. είναι, είναι πολύ περιορισμένα τα πράγματα ερώτηση. Σε ό,τι αφορά όμως ε, τα τελικά αποτελέσματα, σε τελική ανάλυση είναι αντιπροσωπευτικά για το τι συμβαίνει στον δρόμο. Όχι, κοιτάξτε, ο στόχος είναι πάντα το όχημα να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο όχημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί τελικά. Αν χρειάζονται κάποιες αλλαγές προκειμένου να είναι ασφαλή η διεξαγωγή του ελέγχου, όπως για παράδειγμα η πίεση των ελαστικών, νομίζω ότι είναι αποτεκτές αυτές οι τροποποίησεις και η νομοθεσία της ορίζει ξεκάθαρα. Ναι, είμαι περίεργη. Οι υπηρεσίε σας έχουν ποτέ αρνηθεί χορηγήσει τέτοια έγκριση σε κάποιον κατασκευαστή. Κοιτάξτε. Εμείς ε, δίνουμε τα αποτελέσματα των ελέγχων. Είμαστε τεχνική υπηρεσία. Σε κάποιες περιπτώσεις κάναμε ελέγχους και τα οχήματα απέτυχαν και δεν πέρασαν τους ελέγχους αυτούς και χρειάστηκαν να τροποποιηθούν. Εκτός μικροφώνου η ερώτηση. Sorry. Sorry. Have you ever challenged Έχετε ποτέ υποπτευτεί και κατηγορήσει κάποιον κατασκευαστή για το ότι τα οχήματα είναι ανταπροσωπευτικά. Εδώ και τρία χρόνια από την πρώτη σημερινή που δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Πριν από πολλά πολλά παραδείγματα χρόνια ε, είχα ακούσει μια τέτοια περίπτωση για ένα όχημα το οποίο ήταν αμφισβητήσιμο πριν από 20 χρόνια. Δεν είναι κάτι κοινό αυτό γενικά. Σε γενικέ γραμμέ γίνεται επιθεώρηση και διαπιστώνεται ότι τα οχήματα συνάδουν και με την νομοθεσία και με τι προδιαγραφέ. Γενικά οι κατασκευαστέ. ε, Ξέρουμε ποια είναι τα πρότυπα αυτά και δεν ε, αποσκοπούν στο να τα παρακάμψουν. Ο κύριος Γεμπράντη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι τυχερή μου μέρα. Να συζητήσω μαζί σας τον όρο φυσιολογικές συνθήκες χρήσης. Γιατί ήταν κεντρικό θέμα των ερευνών μας αυτό. Στην απάντηση στην ερώτηση περιθμών 9 αναφέρεται ότι οι φυσιολογικές συνθήκες χρήσης δεν ε, ορίζονται επαρκώς. Από την άλλη, από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ίδρυμα για το αναφέρεται ότι πρόκειται για την κανονική χρήση εκτός εργαστριακών συνθήκων. Άρα αυτοί κρίνουν ότι είναι επαρκές. Επαρκής ορισμός του πώς λειτουργεί ένα όχημα εκτός εργαστηρίου. Καταρχάς, ερώτημα απευθυνθήκατε ποτέ τι εθνικέ σα αρχέ για διευκρινήσει σε ό,τι αφορά τον ορισμό αυτό. Κάλεσατε ποτέ τι αρχέ σα να στραφούν προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πιο πολλέ διευκρινήσει. Όχι, κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι το έχουμε, έχουμε ζητήσει σχετικέ διευκρινήσει, αλλά για να είμαστε και ειλικρινεί, αυτό δεν χρειάζεται να μα απασχολήσει και πάρα πολύ. Γιατί ο ρόλο μα στο εργαστήριο είναι να κάνουμε του ελέγχου μέσα στο εργαστήριο και να αναφέρουμε τα αποτελέσματα. Ναι, ναι, ναι, ασφαλώς. Αλλά χορηγείτε και συμβουλές. Δεν βοηθάτε τους, ε, την βιομηχανία να περάσει το τεστ, αλλά τους εξηγείτε τι χρειάζεται για να περάσουν τον έλεγχο για την έγκριση τύπου. Εκεί η ερμηνεία της κανονικής χρήσης ασφαλώς είναι κεντρική. Γιατί αν στο ρόλο σας ως σύμβουλοι τους δηλώσετε ότι τα αρχήματα αυτά θα πρέπει να συνάδουν και με το όρο εκπομπών στο δρόμο, ασφαλώς αυτό είναι πολύ βασικό στοιχείο. Απάντηση. Ναι, κοιτάξτε, πάντα ανατρέχουμε στον κανονισμό και διευκρινίζουμε ότι αυτή είναι η έλεγχη που θα πρέπει να περάσετε για να πάρετε την έγκριση τύπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι, συζητάμε τον ορισμό των ελέγχων ε, με τους πελάτες μας. Όχι το τι είναι η κανονική χρήση. Γιατί η δοκιμή ουσιαστικά πρέπει να αναπαράγει την κανονική χρήση. Άρα αυτό που εξηγούμε στους πελάτες μας είναι τους ελέγχους που θα πρέπει να περάσουν για να πάρουν την έγκριση τύπου. Ναι, γιατί σε τελική ανάλυση το θέμα είναι αυτός ο έλεγχος. Άρα θα πρέπει να αναπτυχθούν το συντομότερο δυνατό αυτή η νέη έλεγχη RDE. Άλλη ερώτηση. Δεν παρέχετε συμβουλές προς του πελάτες σας για το πώ μπορούν να περάσουν πιο εύκολα τους ελέγχους και αυτό πολύ σωστά το κάνετε έτσι. Αλλά φαντάζομαι ότι γνωρίζετε, αντιλαμβάνεστε πόσα πολλά κόλπα μπορούν να γίνουν για να περάσει κανείς πιο εύκολα ένα έλεγχο. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι αυτά τα κόλπα. Τα οποία ενδεχομένω να δώσετε και ως συμβουλή στους πελάτες σας. Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρουμε τέτοια κόλπα για να περάσει κανείς τους ελέγχους αυτούς. Τα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τις δοκιμές παίρνουν από την επιθεώρηση. Υπάρχει πολύ περιορισμένο περιθώριο ελιγμών τροποποίηση των οχημάτων αυτών, όπως σα είπαμε. Και η έλεγχη είναι πολύ ενδέλεχη ω προς τι προδιαγραφέ του. Αν υπάρχει οποιοδήποτε κόλπο, ενδεχομένω να είναι στην κατασκευή του οχήματο. Εκεί δεν ε, μπλεκόμαστε. Κάνουμε και ελέγχους στη φάση της ε, κατασκευής του οχήματος για να κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση ο κατασκευαστής. Κοιτάξτε, αυτό πιστεύω ότι είναι λίγο δύσκολο να το πιστέψω. Δυσκολεύομαι. Γιατί όταν επισκέφτηκα μία από αυτές τις εγκαταστάσεις ε, ελέγχων ήταν σαφές ότι οι τεχνικοί που κάνουν τους ελέγχους ήξεραν τα πάντα, τα μέσα και τα έξω για τα οχήματα αυτά. Όλοι ξέρουμε ο πρώην Επίτροπος Ποτνότσνικ απέστειλε και μία επιστολή προς τον ε, πρώην Επίτροπο Τατσιάνη ότι είναι κοινή γνώση, ότι είναι κοινό στοιχείο. Το ξέρουν όλοι ότι υπάρχουν ε, τέτοιες, τέτοιοι τρόποι για να μας τορέψει κανείς τα οχήματα. Ίσως για σας ε, αυτό να μην αποτελεί καν κόλπο. Να σας το πω κι αλλιώς τα οχήματα τα οποία ελέγχεται για να πάρουν έγκριση τύπου μπορούν αυτόματα να βγουν στον δρόμο. Συμμορφούνται με όλες τις προδιαγραφές που ορίζουμε. Απάντησε. Ναι. Αν υπάρχει μία εξαίρεση, αυτή θα ήταν ενδεχομένω η πίεση των ελαστικών. Είναι πολύ υψηλή για να βγουν στον δρόμο. Και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που γίνονται οι δοκιμέ και οι έλεγχοι στο εργαστήριο. Άρα, ναι, η απάντηση είναι μπορούμε να του βγάλουμε λίγο αέρα και να βγουν στον δρόμο. Good afternoon and thank you for Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Εγώ θα ήθελα να απαντήσουμε στην, ε, να δούμε την απάντησή σας στην ερώτηση 4 που είπατε ότι είδαμε ε, ότι καιρού εις καιρών διαρμηνέθηκαν οι κανονισμοί με διαφορετικό τρόπο ε, και άρα υπήρχαν διαφορετικά αποτελέσματα για συγκεκριμένες πιστοποιήσεις. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ίδιους παραδείγματα είδατε όπου υπήρχαν διαφορετικές ερμηνείες των κανονισμών. Ε, κύριος είναι αυτός ο ορισμός της χειρότερης ε, περίπτωσης αλλά αυτό θα πρέπει να είναι να υπάρχει ένα υποκείμενο εκτίμησης για το είδος των οχημάτων που εντάσσονται στο συγκεκριμένη έγκριση τύπου. Ποιο είναι το όχημα το οποίο έχετε ισχυρότερες εκπομπές, ε, οπότε αυτό δοκιμάζεις. Εάν υπάρχει βεβαιότητα για το ποιο είναι το χειρότερο ή αν θα πρέπει να δούμε δύο, τρία, τέσσερα είναι περίπου όλα ισότιμα και άρα πρέπει όλα να ελεγχθούν. Αυτή είναι η πιο πιθανή περίπτωση και αυτό θα αλλάξει το κόστος αλλά και το χρόνο. Κυρίως το χρόνο που χρειάζεται για να γίνει ένα τεστ έγκριση τύπου. Ναι, πρέπει δηλαδή να ελέγξει κανείς σε τέσσερα διαφορετικά αυτοκίνητα λόγω μιας διαφορετικής ερμηνείας για το τι είναι το χειρότερο αυτοκίνητο. Η έγκριση τύπου καλύπτει πάνω από μία συγκεκριμένη ε, σειρά ε, μοντέλο αυτοκινήτου. Θα πρέπει να αποφασίσουμε λοιπόν ποια μοντέλα θα δοκιμάσουμε κάθε φορά, ώστε να είμαστε αρκετά βέβαιοι ότι όλα τα, τα οχήματα που καλύπτουν από τη συγκεκριμένη έκρηση τύπου αντιστοιχούν και ικανοποιούν τους κανονισμούς. Είδατε οι αρχές ε, να ζητούν περισσότερους ελέγχους, αλλά λιγότερους ε, ελέγχους τύπου, εγκρίσεις τύπου. Όχι, δεν έχω στοιχεία για να πω κάτι τέτοιο. Δεν, έχω να, δεν μπορώ να πω. Θα πρέπει να ρωτήσετε τους κατασκευαστές των αυτοκινήτων γιατί επιλέγουν τη συγκεκριμένη αρχή έγκρισης τύπου. Συχνά αυτό οφείλεται στην εγκύτητα και συχνά οφείλεται στο χρόνο που παίρνει μια τέτοια έγκριση τύπου γιατί θέλουν να βάλουν τα προϊόντα στην αγορά, να κυκλοφορήσουν τα προϊόντα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Του ρωτήσαμε, του κατασκευαστέ, αλλά δεν ε, μα τα είπαν και πολύ ξεκάθαρα. Και πράγμα το οποίο δεν μα εξέπληξε βέβαια και τόσο. Τώρα, όταν με, μιλήσαμε με συναδέλφους σας ε, για τη Γερμανία είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα στάνταρ για το χρυσό αυτοκίνητο, χρυσό κανόνα ας πούμε για τα αυτοκίνητα. Ε, μπορείτε εσείς να μας εξηγήσετε ποιος ορίζει τις ε, παραμέτρους για τα, τις δοκιμές. Ε, μάλλον είδατε το τεστ αυτό ε, στο, εργασ... στο εργαστήριο στη διάρκεια του, της δοκιμής close down. Ε, ποιος κάνει αυτές τις δοκιμές. Υπάρχουν άλλες ε, εγκαταστάσεις για δοκιμές ε, κατάλληλες για αυτό το ίδιο. Υπάρχει ένα τέτοιο, ε, σε τέτοιο, μια τέτοια κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο καιρό είναι αρκετά μεταβλητός, έχουμε 6 χιλιόμετρα διαδρομή είναι ευκολότερο να γίνει τέτοιο τεστ close down σε, μακρύτερο, σε μακρύτερη διαδρομή. Γι' αυτό και οι κατασκευαστές συνήθως πηγαίνουν σε άλλα μέρη στην Ευρώπη, ή στις ΗΠΑ, όπου ο καιρός είναι πιο αξιόπιστος Τι θα πει αξιόπιστο, αξιόπιστο που θα πει που δίνει καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί για να σα πω ειλικρινά, αυτό που ακούσαμε είναι ότι τελικά οι κατασκευαστέ παίρνουν αυτέ τι παραμέτρου του test close down και μετά εσεί ω ως ε, ε, στοιχείο της δοκιμασίας παίρνετε αυτά τα στοιχεία. Παίρνετε αυτά τα στοιχεία από τα test close down. Από τους κατασκευαστές δηλαδή. Όχι, γιατί τα close down είναι κομμάτι της έγκρισης τύπου. Είναι το ίδιο σημαντικά με τα δοκιμές για τις εκπομπές και θα πρέπει να γίνονται υπό τις ίδιες συνθήκες εποπτείας όπως και οι δοκιμές για τις εκπομπές. Θα πρέπει να γίνονται από εργαστήρια εγκεκριμένα υπό την εποπτεία τεχνικής υπηρεσίας που με τη σειρά της εποπτεύεται από την αρχή έγκρισης τύπου. Το close down λοιπόν είναι κομμάτι της έγκρισης τύπου. Και ποιος είναι ο αντίκτυπος, γιατί ξέρουμε ότι αυτές οι παράμετροι μπορεί να καθοριστούν εξ αρχής. Ποιος είναι ο πιθανός αντίκτυπος στα δικά σας αποτελέσματα, ανάλογα με τις διαφορετικές παραμέτρους επί τη βάση των δοκιμών close down. Κοιτάξτε, τα αποτελέσματα αυτά έχουν αντίκτυπο στο τεστ ε, εκπομπών, αλλά τι αντίκτυπο. Είπατε ότι υπάρχουν διαφορετικές παράμετροι, άρα ξέρετε περίπου ποιος είναι ο αντίκτυπος. Όχι. Εμείς γνωρίζουμε τις, ε, παραμέτρου, τις, ε, τα αποτελέσματα close down που έχουμε κάνει εμείς οι ίδιοι τις δοκιμές ή που μας δίνονται δεν, αλλά δεν ξέρω ποια είναι η αναλογία. Ποια είναι η διαφορά. Εάν οι δοκιμές close down γίνονται με συγκεκριμένο πάντα ίδιο τύπο, ε, τότε ο αντίκτυπος ε, σε εκπομπές δεν είναι τόσο μεγάλος. Ναι, αλλά αυτές οι παράμετροι δεν είναι πάντοτε πραγματικές συνθήκες. Ε, κοιτάξτε, οι αρμόδιοι για την εποπτεία της αγοράς είναι αυτοί που κάνουν ε, τις δοκιμές ε, επιτόπου σε πραγματικές συνθήκες, θα πρέπει να μπορούν να σας πούν. Κυρία Εύη, ευχαριστώ. Εγώ έρχομαι εκ νέου στο θέμα του χρυσό κανόνα για το αυτοκίνητα, γιατί σύμφωνα με μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Περιβάλλον, ο οργανισμός δείχνει 8 διαφορετικές ε, δοκιμές ένα το αναφέραμε ε, για τα ελαστικά, ας πούμε, αλλά και για το ε, ειδικά λιπαντικά έλαια και ούτω καθεξής, ανάλογα με τις δοκιμές, διαφορετικά το κόλπα δηλαδή. Θέλω να ξέρω κατά πόσο αυτές οι ενδείξεις είναι αληθινές, γιατί εδώ θέλουμε να καταλάβουμε ποιος λέει ψέματα. Αν ε, όντως, αν υπάρχουν δηλαδή αυτά τα χρυσά αυτοκίνητα ή όχι. Εμείς ε, θα πρέπει να σας πω ότι δεν έχουμε κάποιο δίκτυο για τέτοια χρυσά αυτοκίνητα. Δεν ξέρω ποια είναι τα χαρακτηριστικά που επιλέγουν οι κατασκευαστές για να περάσουν ένα αυτοκίνητο από το ε, ναι, δοκιμή έγκρισης τύπου ε, το εξάλλου η δοκιμή ελέγχου εποπτείας της αγοράς που θα γίνει στο μέλλον θα δείξει σημαντικές διαφορές σε σχέση με το δοκιμή που κάνουμε εμείς υπό την έγκριση τύπου και έπειτα η αρχή έγκριση τύπου θα πρέπει να ερευνήσει το λόγο στον οποίο οφείλεται αυτή η διαφορά. Και εφόσον κανεί χρησιμοποιεί το χρυσό αυτοκίνητο για να επιτύχει σημαντική μείωση των εκπομπών στη διάρκεια των δοκιμών για την έγκριση τύπου, θα φανεί αυτό στα αποτελέσματα της ε, εποπτείας της αγοράς. Ναι, μάλιστα. Ευχαριστώ. Είναι λυπηρό να χρησιμοποιούμε ακόμα ότι θα φανεί και ότι θα γίνει, γιατί δυστυχώς το συζητάμε εδώ και πολύ καιρό και γνωρίζουμε το τι συμβαίνει εδώ και αρκετό καιρό. Τώρα, σύμφωνα με την δική σας άποψη, είπατε ότι το μοντέλο της πιστοποίησης θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο παρόμοιο, πιο ίδιο με το αυτοκίνητο που βγαίνει από την παραγωγή. Αν ε, συγκεντρώσουμε τις διάφορες μικροδιαφορές ανάμεσα στο μοντέλο που πιστοποιείται και τα αυτοκίνητα που βγαίνουν από την αλυσίδα παραγωγής, τι ποσοστό απόκλησης θα μπορούσατε να μας δώσετε ότι υπάρχει.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 δεν μπορώ να το ποσοστοποιήσω. Απλά θα πρέπει να διευκρινίσω ότι στο μέλλον, έτσι όπως σήμερα είναι συνταγμένος ο κανονισμός και όπως ισχύει εδώ και αρκετά χρόνια, είναι το εξή ισχύει. Ότι δηλαδή υποβάλλεται στην έγκριση τύπου ένα αυτοκίνητο και μετά γίνεται υποπτή αγορά στα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην αγορά. Και αυτό γίνεται μετά από την έγκριση τύπου. Αλλά αυτό θα γίνεται και στο μέλλον. Είναι κάτι που θα έπρεπε να γίνεται και σήμερα κανονικά. Μάλιστα. Σα ευχαριστώ. Μια τελευταία ερώτηση. Σύμφωνα με τη δική σας κρίση, το βασικό αίτιο για τα ψηλά επίπεδα εκπομπών οξυδίων του αζότου στην ατμόσφαιρα ε, οφείλεται κυρίως στη χρήση παράνομου λογισμικού, δηλαδή συσκευών αναστολής ή στην ιδέα ότι μπορούν να πιστοποιούνται αυτοκίνητα τα οποία σέβονται τα όρια μόνο και αποκλειστικά στο εργαστήριο και άρα υπάρχουν σοβαρές διαφορές ανάμεσα στη μέσα στο εργαστήριο και στην πραγματικότητα. Πιστεύω ότι το τελευταίο ισχύει γιατί νομίζω πως η ανάπτυξη των αυτοκινήτων, η εξέλιξη μάλλον των αυτοκινήτων έχει περάσει σε πολύ διαφορετικό επίπεδο. Χρησιμοποιούνται τα αυτοκίνητα με πολύ διαφορετικούς τρόπους από ότι ο κύκλος που έχει αναπτυχθεί για αυτή την έγκριση τύπου και ο κανονισμός δεν έχει ε, συμβαδίσει με την ανάπτυξη των αυτοκινήτων, την εξέλιξη μάλλον των αυτοκινήτων και αυτό είναι το πρόβλημα το βασικό. Οι εκπομπές ε, δηλαδή που μετρώνται στη διάρκεια αυτών των δοκιμών δεν είναι ίδιες με αυτές που είναι, γίνονται στην πραγματική χρήση. Συγγνώμη, καθυστέρησα σε μια άλλη συνεδρίαση. Η Μίλμπροκ ε, έχει ε, δύο συστήματα, ε, φορητά συστήματα μέτρησης καταλήγει σε ένα δείκτη συμμόρφωση 2,1. Πώς καταλήγει αυτό και από τεχνικής πλευράς είναι οι καλύτερες μετρήσεις που μπορούμε να κάνουμε. Τι συμβουλή θα μας δίνατε εμάς, τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε το σύστημα έγκρισης τύπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι κατά την άποψή σα για το σκάνδαλο των εκπομπών από πλευρά διαδικασίας έγκρισης τύπου αλλά... Να απαντήσω μία-μία τις ερωτήσεις σας. Χρησιμοποιούμε PEMS, φορητά συστήματα μέτρης καυσέρων εδώ και δύο-τρία χρόνια. Ε, αργά ε, στην αρχή, αλλά όλο και περισσότερο προϊόντος του χρόνου. Ε, οι κατασκευαστές δυσκολεύονται να βρουν καλές τέτοιου τύπου διατάξεις συσκευές PEMS ε, σιγά σιγά ε, υπάρχουν όλο και καλύτερες στην αγορά. Πιστεύουμε ότι είναι αρκετά ακριβής πια. Ε, ε χρησιμοποιούμε άλλου τύπου συσκευές για να συγκρίνουμε με τα αποτελέσματα των PEMS. υπάρχει μια απόκληση, αλλά πάντως δεν είναι πολύ μεγάλη. Πιστεύω ότι ο παράγοντας συμμορφωσης 2,1 ε, είναι αρκετά πολύ περιοριστικός και αυστηρός για τους κατασκευαστές. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι η τα καυσαέρια, οι πομπές κατά τη χρήση είναι 5 6 φορές περισσότερα. Η μείωση του 6 στο 2,1 είναι ένας πολύ δύσκολος στόχος για τους κατασκευαστές. και νομίζω ότι αφιερώνουν πολύ προσπάθεια και χρόνο αυτή τη στιγμή για να το καταφέρουν. Σε ό,τι αφορά την τροποποίηση των κανόνων και της νομοθεσίας προκειμένου να αποφύγουμε αυτή την αύξηση της διαφοράς ανάμεσα στις αραστηριακές δοκιμές και στην πραγματικότητα ε, νομίζω ότι για να το πετύχουμε χρειάζεται μια ε, ένα, μια, επαρκή ποικιλία συνθήκων ε, στις πραγματικές δοκιμές επιτάχυνσης, ταχύτητας και θερμοκρασίας για παράδειγμα που να, να αντιπροσωπεύουν τι πραγματικά συμβαίνει ε, όταν οι οδηγοί χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους και βέβαια ένας παράγοντας συμμόρφωσης που θα έχει ε, θα, έχει, θα είναι λογικός ε, σε ό,τι αφορά το τι μπορούμε να περιμένουμε από τους κατασκευαστές στο μέλλον σε σχέση με αυτό που έχουμε σήμερα. Ευχαριστώ. Περνάμε στον επόμενο γύρο ερωτήσεων. Κύριο Σούλτσε. Ε, um, Κύριε Μπέρνς, σας ευχαριστώ και από δικής μου πλευράς. Σας ευχαριστώ και εγώ για Ήθελα να αναφερθώ στην υφιστάμενη νομοθεσία. Όλοι ομολογούν ότι έχει αδυναμίες. Και οι αδυναμίες αυτές εντοπίζονται από όλους όσους έχουν έλθει τώρα στην Επιτροπή μας. Αυτό που θα ήθελα να μάθω είναι το εξής. Τα τελευταία χρόνια πώς έχει διαμορφωθεί η επικοινωνία σας με τις βρετανικές αρχές και με τις κοινωτικές αρχές σε περίπτωση αδυναμιών, σε περίπτωση προβλημάτων. Ενημερώνατε. Ή θεωρείτε ότι η νομοθεσία έχει ως έχει και εσείς απλά την εκτελείτε και δεν μπλέκεστε σε περαιτέρω απόπηρεσία για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Σας ευχαριστώ στον Ηνωμένο Βασίλειο ε, συνεισφέρουμε και εμείς τις συζητήσεις για το τι μορφή θα πρέπει να πάρουν στο μέλλον η, να πάρει στο μέλλον η κανονιστική, το κανονιστικό πλαίσιο ε, και οι εκπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου προωθούν αυτές τις απόψεις. Ε, είμαστε γενικά υπέρ της επικαιροποίησης των κανονισμών έτσι ώστε οι κύκλοι δοκιμής να εξυγχρονιστούν. Όπως και πολλοί άλλοι πιστεύουμε ότι ο νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης, ο NEDC, έχει ξεπεραστεί και θα πρέπει να επικαιροποιηθεί. Από εμπορική πλευρά, ε, είμαστε υπέρ κανόνων που απαιτούν περισσότερες δοκιμές. Ε, εν γέννη προσπαθούμε να υποστηρίξουμε μια υγιή αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη. Οπότε η δική μας συνεισφορά είναι μέσω διαβημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο υπέρ της ε, μετακίνησης προς την ε, ε, RDE, προς, τον, προς τις διαδικασίες μέτρησης πραγματικών εκπομπών, την WLDP κλπ. Θέλουμε δηλαδή να οθήσουμε την αυτοκινητοβιομηχανία σε μια υγιή κατάσταση. Σας ευχαριστώ και μιας και δείξατε το θέμα των διατάξεων ελέγχου και δοκιμών να αναφερθώ σε κάτι άλλο. Είσαστε σε θέση ή είσαστε σε θέση να διεξαγάγετε τους ελέγχους αυτούς μόνο στις δικές σας εγκαταστάσεις ή μήπως αναγκαστήκατε σε διάφορες περιστάσεις να κάνετε και τέτοιες δοκιμές στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Εμείς ε, λειτουργούμε ως εργαστήριο, οπότε οι δοκιμές γίνονται στις δικές μας εγκαταστάσεις. Ε, οι δοκιμές εκπομπών ε, είναι είναι μια δραστηριότητά μας από το 1970. Ε, οπότε οι εγκαταστάσεις μας στο εργαστήριο μας είναι σχετικά παλιό. Σκοπεύουμε να χτίσουμε, να δημιουργήσουμε ένα καινούριο εργαστήριο ε, που ε, θα ε, είναι προσαρμοσμένο στο νέο κύκλο και θα βοηθήσουμε αυτόν τον τρόπο την βιομηχανία στο να προσαρμοστεί καλύτερα στην κοινωνική πραγματικότητα. Επίσης επενδύουμε σε φορητές ε, διατάξεις με τι καυσέριων, PEMS, καθώς επίσης και σε ε, δημιουργία ε, εγκεκριμένων πιστών, εγκεκριμένες πίστες για μέτρηση καυσαρίων σε πραγματικέ συνθήκες. Θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να έχουμε ένα, ε, ε, θα πρέπει να έχουμε ένα περιβάλλον δικό μας, ιδιωτικό περιβάλλον ε, δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες έτσι ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την καινούργια διαδικασία RD. Ευχαριστώ κύριε Μπέρν που είστε εδώ μαζί μας. Μας είπατε ότι ήταν μεγάλη έκπληξη για σας όταν έσκασε το σκάνδαλο. Φαντάζομαι όμως ότι έχετε πολλούς τεχνικούς και πολλούς ε, ε, μηχανικούς στην εταιρεία σας και ξέρουν τα πάντα για τις δοκιμές. Ε, προφανώς δεν είναι δικό σας φάλμα, αλλά αναρωτιέμαι πώς είναι να το κάνεις πουθενά να μην είχε υποψίες για το γεγονός ότι μια εταιρεία θα μπορούσε να εξαπατήσει τις αρχές και το κοινό με τη χρήση τέτοιων ε, διατάξεων Ήδη στι ΗΠΑ από το 1998 ξέρουμε ότι υπήρχαν εταιρείε που είχαν τέτοιου διατάξει. Ε, Πώ είναι δυνατόν να σα εκπλήσει τόσο πολύ ότι μια εταιρεία μπορεί να θέλει να εξαπατήσει. Ε, δεν με εξέπληξε, εγώ είπα σοκαρίστηκα. Ε, Ήταν ε, πολύ πιο έντονο. Ε, ε, και ήταν έτσι γιατί σύμφωνα με τη δική μας εμπειρία. Οι κατασκευαστές εργάζονται πάρα πολύ σκληρά για να τηρήσουν την νομοθεσία και τους κανόνες και κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου τα αυτοκίνητα τα οποία εμπορεύονται να συμμορφώνονται με τους κανόνες πάντα. Βέβαια, γνωρίζαμε την όλο και μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στις εργαστηριακές δοκιμές και στην πραγματικότητα, την οποία εμείς, όπως σας είπα και προηγουμένως, αποδίδαμε ε, στην ταχεία εξέλιξη των οχημάτων. Όμως, ερώτηση, όμως εσείς την εταιρεία σας εσωτερικά συζητούσατε ποτέ ε, την πιθανότητα αυτή να οφείλεται σε τέτοιες διατάξεις αναστολής. Ε, γενικά λέγαμε ότι αυτή η διαφορά οφείλεται στο γεγονό ότι ο κύκλος δοκιμών είναι πεπαλαιωμένος, ξεπερασμένος και δεν παρακολουθούσε την, εξελίξει στην ε, παραγωγή των αυτοκινήτων. Οπότε είχαμε την εντύπωση ότι τα αυτοκίνητα είναι νόμιμα, απλά εξελίσσονται τεχνολογικά πολύ γρήγορα. Ωραία, αυτό είναι το παρελθόν. Τώρα έχουμε καινούργια νομοθεσία που προσπαθεί να βελτιώσει την πρόταση της Κομισιόν. Θέλω να βρούμε έναν τρόπο για να αλλάξουμε την οτροπία και τον τρόπο σκέψης τόσο των νομοθέτη όσο και των κατασκευαστών. Πώς μπορούμε να χτίσουμε μέσα στο σύστημα, να εντάξουμε στο σύστημα περισσότερες υποψίες, να το κάνουμε πιο φιλίποπτο. Ε, όταν υπάρχουν υπόνοιες, ε, να αντιδρούμε πιο εύκολα, πιο γρήγορα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό μέσα της νομοθεσίας κατά την άποψή σας. Απάντηση. Ορισμένα από αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή ε, με τις διαδικασίες RDE και WLTP είναι καλά. Ε, η, επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε την υποπτία της αγοράς. Ήδη φύστανται κανόνες για την υποπτία της αγοράς, αλλά ενδεχομένω δεν είναι επαρκής η υποπτία αυτή τη στιγμή. Από την άλλη μεριά η εποπτεία της αγοράς είναι ο μηχανισμός ο οποίος ε, ε θα απέτρεπε, θα δρούσε ως αποτροπή έναντι ε, τέτοιων προσπαθειών ε, παραποίησης. Ε, αν ο κίνδυνος σε μεγάλο σε πιάσουν θα το αποφύγεις. Ερώτηση. Είχαμε την EPA εδώ πριν από μερικές εβδομάδες και μας είπαν ότι έχουν προσθέσει πλέον ένα στοιχείο ε, μη προβλεψιμότητας στις ε, δοκιμές. Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο είναι καλό. Ναι, το διάβασα και εγώ και ρώτησα τους μηχανικούς μου τι σημαίνει αυτό και ούτε οι μηχανικοί μου ξέρανε. <laughs> Με λείψε βέβαια πολύ αυτό. Πρέπει να υπάρχουν όμως και όρια σε αυτό. Γιατί ε, σκεφτείτε ότι είστε ε, κατασκευαστής. Προσπαθείτε να αναπτύξετε ένα αυτοκίνητο που να τηρεί συγκεκριμένου κανόνες. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια. Γιατί αν πάρετε ένα πολύ κρύο αυτοκίνητο και το επιταχύνετε από τους πρόποδες των άλπων μέχρι την κορυφή, ε, θα εκπέμψει πάρα πολλά καυσαέρια, πολλούς ρήπους. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον κατασκευαστή ότι ε, ε, δεν θα πρέπει το αυτοκίνημα του να ξεπερνάει τα όρια. Οι Συνωμένες Πολιτείες όμως έχουν το νόμο Cleaner, Cleaner Act. Ε, και τα αυτοκίνητα, οι μηχανίες πρέπει να συμμορφώνονται. Εμείς εδώ έχουμε την έγκριση τύπου. Μήπως θα πρέπει και εμείς να πούμε ότι ο βασικός μας στόχος είναι ο καθαρός ο ατμοσφαιρικός αέρας και τίποτα άλλο. Απάντηση. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και στα δύο συστήματα και στις δύο προσεγγίσεις. Το αμερικανικό σύστημα ε, ε, μεταφέρει ένα μεγάλο τμήμα της ευθύνη στους κατασκευαστές και μετά ε, επιβάλλει ευστήρα πρόστιμα αν αυτοί δεν τα καταφέρουν να συμμορφωθούν. Το μειονέκτημα αυτού είναι ότι ε, μπορεί να ε, δημιουργήσει μια ε, ασάφεια σε ό,τι αφορά το ποιοι είναι κανόνες με τους οποίους πρέπει να συμμορφωθούν οι κατασκευαστές. Και αυτό ενδεχομένως δεν βοηθάει πολύ την ανάπτυξη καινούργιων αυτοκινήτων. Το ευρωπαϊκό σύστημα λέει πρέπει να περάσει αυτά τα ε, τεστ, αυτές τις δοκιμές και αν η εποπτεία της αγοράς ε, είναι επαρκής, θα μπορέσουμε μάλιστα να διαπιστώσουμε και να διαπιστώνουμε συνεχώς αν τα αυτοκίνητα συνεχώς συμμορφώνονται. Μήπω θα μπορούσαμε όμω να πάρουμε τα καλά στοιχεία του Αμερικανικού συστήματο και να τα μεταφέρουμε σε εμά, γιατί αυτοί εντόπισαν το σκάνδαλο, ε, δεν το ανακαλύψαμε εμεί. Αν δείτε ε, το εύρος των κύκλων που χρησιμοποιούν, ε, θα δείτε ότι μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Ε, δεν καταλαβαίνω μάλιστα και τον παράγοντα μη προβλεψιμότητας. Ε, αν δεν ξέρουν οι κατασκευαστέ ποιε είναι οι διαδικασίε, πώ θα συμμορφώνουν τα οχήματά του. Μήπω όμω θα ήταν καλό για του πολίτε και την υγεία. Ναι, το καταλαβαίνω. Και ασφαλώς είναι επιθυμητό. Αλλά θέλετε, θέλουμε οι, κανονισμοί να γίνονται αντιληπτοί από αυτούς που θα τους εφαρμόσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Μπέρνς, ε, ήταν ενδιαφέρον ε, το απόγευμα και ενδιαφέρουσα και δήλωση ότι σοκαριστήκατε αλλά δεν εκπλαγήκατε. Δηλαδή πώς έγινε αυτό το πράγμα, σοκαριστήκατε αλλά δεν εκπλαγήκατε. Τι να σας πω, καλό μάθημα για τους βουλευτές αυτό σε ό,τι αφορά τα θέματα ανεξαρτησία τώρα. Στη γράπτη σα απάντησε στην ερώτηση παριθμών 5 απαντάτε στην κατηγορία ότι υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων όταν η Μίλμπροκ ακόμα ανήκε στην General Motors και τονίζετε ότι έχετε προσωπικό υψηλή εξειδίκευση. Μπορείτε να μου πείτε πόσους εμπειρογνώμονες ε, έχετε από την αυτοκινητοβιομηχανία ή πόσοι από τους εμπειρογνώμονές σας μετά την απασχόληση στην εταιρεία σας πηγαίνουν στην ε, αυτοκινητοβιομηχανία. Απάντηση, κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές οι υπάλληλοι μας έχουν ε, δουλέψει στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην βιομηχανία διεξαγωγής ελέγχων κτλ. Είναι από μέσα από την ε, βιομηχανία για το μεγαλύτερο μέλος, μέρος της καριέρας τους. Υπάρχει λοιπόν τεχνική εμπειρογνωμοσύνη. Δεν ξέρω, απαντήθηκε έτσι η ερώτησή σας. Το ερώτημα είναι κατά πόσον υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων αν ένας πρώην υπάλληλος της General Motors τώρα κάνει υποπτία σε οχήματα General Motors στην πολιτική υπάρχει περίοδος εξαίρεσης και δεν ξέρω αν υπάρχουν εσωτερικοί κανόνες για τους υπαλλήλους που προέρχονται από κάποια εταιρεία οι οποίοι ενδεχομένω να μην έχουν δυνατότητα να ελέγχουν τα οχήματα της συγκεκριμένη εταιρεία. Υπάρχει κάτι τέτοιο. Όχι, δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες. Οι κανόνες που υπάρχουν είναι ότι αναφέρουμε τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από τις δοκιμές οι οποίες είναι υψηλών προδιαγραφών σχεδόν όλοι οι εταιροί, οι μας ήταν, απασχολούνταν από τη Μίλμπρουκ, γιατί ήταν το τμήμα της ε, General Motors. Λίγοι λοιπόν είναι αυτοί που δεν είναι υπάλληλοι της ε, GM. Ωστόσο έχουμε συστήματα ποιότητα, τα οποία εφαρμόζουμε, γίνεται εξωτερικό έλεγχο και ένα εργαστήριο το οποίο το παρακολουθούν οι τεχνικές υπηρεσίες. Υπάρχουν λοιπόν πολλές τεκλίδες ασφαλείας οι οποίες εξασφαλίζουν ότι αναφέρουμε μόνο τα πραγματικά αποτελέσματα και είναι βασικό στοιχείο, θεμελιώδης στοιχείο για την ε, υγιεινή, αν θέλετε, και την υγεία της υπηρεσίας μας, του οργανισμού μας, το να δρούμε ανεξάρτητα. Μία άλλη ερώτηση, κύριε να αναφερθώ στην απάντηση του Ιταλού συναδέλφου, δεν ξέρω αν ήσασταν εδώ, ο οποίος ε, δήλωσε ότι το σύστημα ανακυκλοφορίας καυσαρίων απονεργοποιείται μετά από 22 λεπτά και ότι αυτό υποτιθέμενα προστατεύει τον κινητήρα. Με την τεχνική σας γνώση, πώς αξιολογείτε αυτή τη δήλωση. Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να το σχολιάσω γιατί δεν είμαι μηχανικός. Δεν έχω προσωπικά την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για να καλύψω το θέμα αυτό. Θεωρώ ότι αυτό θα ήταν αποδεκτό μόνο αν ο κατασκευαστής πραγματικά είχε πείσει τις αρχές χορήγησης έγκρισης τύπου ότι χρειαζόταν αυτή η επινεργοποίηση για την προστασία του κινητήρα. ερώτηση. Μάλιστα. Άρα θα περιμένω την απάντηση της τεχνικής σας υπηρεσίας, γιατί το ερώτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ίσως θα μπορούσατε να μας απαντήσετε για την ε, συνεργασία μεταξύ εργαστηριών. Ας μην λάβουμε υπόψη το Brexit. Θέλετε να φύγετε από την ε, ωραία και όμορφη Ευρωπαϊκή μας Ένωση. Υπάρχει όμως κάποια συνεργασία με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες ή δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Αν γίνεται, πιστεύετε ότι υπάρχει ανταγωνιστικότητα με τα, μεταξύ εργαστηρίων. Απάντηση. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ε, και εγώ νομίζω ότι είμαι τόσο θλιμμένος για τον Brexit τόσο και εσείς. Σε ό,τι αφορά τα εργαστήρια, σε κάποιο επίπεδο ασφαλώ υπάρχει ένα ανταγωνισμό γιατί υπάρχει μια ανάλογη υπηρεσία την οποία παρέχουμε. Αλλά όπω σε πολλέ περιπτώσει ανταγωνισμού έχουμε κοινά συμφέροντα. Το κοινό συμφέρον είναι η επιβίωση του κλάδου και η υγεία του κλάδου. Και εκεί πρέπει να σας πω ότι συνενωνόμαστε σε συνδικάτα, σε φόρουμ βιομηχανικά, όπου συζητούμε την έγκριση νέων κανονισμών και εξασφαλίζουμε ότι ως ε, βιομηχανία, ως κλάδος, είμαστε όλοι συντανισμένοι για να παρέχουμε τις υπηρεσίες δοκίμης και ελέγχου που ζητούν οι πελάτες μας. Άρα θεωρώ ότι είμαστε ένα τμήμα του συνολικού μείγματος του καθορισμού του τι τεστ θα πρέπει να γίνονται, πότε και κατά πόσον η βιομηχανία ανταποκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Η πρόεδρος, επόμενος ομιλητής. Σας ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Μπάρνς για τις σαφείς του απαντήσεις. Έχω ένα μικρό πρόβλημα. Ε, εγώ Είχα κάνει μια σειρά από ερωτήσει, προετοιμάσει μάλλον, αλλά στη διάρκεια τη συζήτηση σιγά σιγά ετέθησαν. Γι' αυτό θα κάνω πιο απλέ ερωτήσει. Η πρώτη είναι η εξή. Υπάρχουν συμπεριφαρέ συγκεκριμένε που υιοθετούν οι κατασκευαστέ αυτοκινήτων που μπορούν κατά κάποιο τρόπο να οριστούν ως συσκευές αναστολής. Για παράδειγμα, το να σταματά ο έλεγχος των εκπομπών κάτω από τους 17 βαθμούς και επειδή προηγουμένως έγινε αναφορά στις θερμοκρασίες των κινητήρων. Στην συζήτηση που έχουμε κάνει μέχρι τώρα ακούσαμε ότι οι εκπομπές είναι περισσότερες όταν γίνεται θερμοεκκίνηση. Αυτό δεν είναι αντίθετο με την ε, λογική ότι δηλαδή ένας κινητήρας που είναι ήδη θερμός ε, θα έπρεπε να έχει φτάσει σε ένα επίπεδο εκπομπών πιο σταθερό και άρα να μην αυξάνονται περισσότερο ακόμα οι εκπομπές. Για το πρώτο κομμάτι της ερώτησής σας. Δεν έχουμε αποδείξεις ε, στις δικές μας δοκιμές ε, για, την, για χρήση των συσκευών αναστολής και γι' αυτό και σοκαριστήκαμε όταν ξέσπασε το σκάνδαλο της Volkswagen. Ξέρουμε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις μετρήσεις στο δρόμο, σε πραγματικές συνθήκες και τις μετρήσεις εν δύση. Αλλά εμείς δεν είδαμε αποδείξεις στις δικές μας δοκιμές για ύπαρξη μηχανισμών αναστολής. Όσον αφορά την θερμό εκκίνηση ή την ψυχρό εκκίνηση, να σας πω ότι καταρχάς ότι εγώ δεν είμαι ο ίδιος μηχανισμός, αλλά σίγουρα τίθεται ερώτημα. Εάν υπήρχαν τέτοιου είδους ενδείξεις, ότι δηλαδή η ψυχρό εκκίνηση δίνει καλύτερα αποτελέσματα από την ενθερμό. Αυτό μηχανικοί θα πρέπει να το εξηγήσουν αν, και εφόσον ισχύει. Σας ευχαριστώ. Έχω μια άλλη γρήγορη ερώτηση που θέλω να σας θέσω. Σίγουρα στη διάρκεια αυτών των ακροάσεων ακούσαμε σιγά, ανακαλύψαμε σιγά σιγά πόσο περίπλοκο είναι το σύστημα των ελέγχων και πόσο περίπλοκος είναι και ο μηχανισμός ε, των ελέγχων. Ε, και γι' αυτό και κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι εντυπωσιακό είναι ότι συχνά χρησιμοποιούνται τα εργαστήρια των ίδιων των κατασκευαστών αυτοκινήτων για να γίνουν οι δοκιμές που στόχο έχουν να ελέγξουν τις εκπομπές. Βρίσκω και ρωτώ τη γνώμη σας, πιστεύω ότι είναι αντιφατική αυτή η υπόθεση. Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων να στρέφεται κανείς δηλαδή στα εργαστήρια μιας εταιρείας η οποία στην ουσία ελέγχεται για τις εκπομπές της. Um, ναι, ως επαγγελματίες μπορώ να σας πω πως είναι δυνατόν για επαγγελματίες που δουλεύουν με ακαιρεότητα να κάνουν τεστ, να κάνουν δοκιμές και να επικυρώνουν την εργασία συναδέλφων στην ίδια εταιρεία. Εγώ αρχικά εργαστήκα στην αεροναυπηγική και το ίδιο γίνεται και εκεί. Ήμουν μάλιστα μάνατζερ ποιότητας. Ε, για αρκετά χρόνια. Ποτέ δεν είχε δημιουργηθεί πρόβλημα για να χρειαστεί να ελεγχθώ εγώ για τα προϊόντα τα οποία τοποθετούνταν πάνω σε αεροσκάφη, τα οποία μάλιστα συχνά οδηγούσα και εγώ ίδιος ως πιλότος. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα λοιπόν. Υπάρχει σύστημα ασφαλιστικών δικλείδων, ώστε εάν κάποιος κατασκευαστής και το εργαστήριό του χρησιμοποιείται ως ε, δοκιμαστικό εργαστήριο, τότε το ο έλεγχο που γίνεται εκεί θα πρέπει να εποπτεύεται από την τεχνική υπηρεσία και από τη στιγμή που υπάρχει ανεξαρτησία ανάμεσα την τεχνική υπηρεσία και το εργαστήριο, όποιο και αν είναι αυτό το εργαστήριο, δεν θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα. Η πρόκληση φυσικά είναι το να το καταλάβουν αυτό οι καταναλωτέ σε αυτήν εδώ την περίσταση. Αυτό είναι ε, θέμα επικοινωνιακό όμω. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Σάλμπα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Μπάρνς, θα ήθελα να, να επιστρέψω στα... σε ερωτήσεις που υπέβαλε ο κύριος Εκχότ σε σχέση με τις διαφορές ερμηνείας ε, στην ε, στις δοκιμές πιστοποίησης. Εσείς θεωρείτε πως υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στις διαφορές αυτές ερμηνείας και τις υποθε... περιπτώσεις ε, χωρών όπως το Λουξεμβούργο που δεν υπάρχει κατασκευαστή αυτοκινήτων αλλά Ε, προστρέχουν σε αυτό πολύ για την ε, επικύρωση ε, και την πιστοποίηση ή το Ηνωμένο Βασίλειο που έχει πολλούς κατασκευαστές αυτοκινήτων και γίνονται αλλού οι πιστοποίησεις. Δεν ξέρω ακριβώ και αν και κατά πόσο οι κατασκευαστέ του Ηνωμένου Βασιλείου πηγαίνουν αλλού για πιστοποίησεις. Δεν είδα κανένα να πηγαίνει στο Λουξεμβούργο εγώ ίδιο. Οπότε καλύτερα είναι να του ρωτήσετε εκείνου. Νομίζω πω μάλλον πρέπει να έχει να κάνει με το χρόνο, γιατί περισσότεροι με το χρόνο έχουν να ασχοληθούν, γιατί ο χρόνος είναι βασικός παράγοντας ε, κριτήριο μάλλον για τους κατασκευαστές. Έχω δει ένα παράδειγμα ενός κατασκευαστή λεωφορείου, λεωφορείων ε, που χρησιμοποιεί ως κριτήριο το κόστος, αλλά είναι ένας. Περισσότεροι εξετάζουν το πόσο γρήγορα θα μπορέσουν να πιστοποιήσουν το προϊόν τους, ώστε να χρησιμοποιηθεί και να μπει στην αγορά γρήγορα. Μάλιστα. Από τα όσα είπατε λοιπόν κατανοώ ότι αυτή η διαφορετική ερμηνεία που αναφέρεται στη γραπτή σας απάντηση δεν σχετίζεται με τη χώρα στην οποία γίνεται η πιστοποίηση, εκεί που χρησιμοποιείται περισσότερο. Για παράδειγμα, χειρότερη ε, το χειρότερο παράδειγμα που σας έδωσα και νωρίτερα είναι ότι αν μία αρχή έγκρισης τύπου ζητά πολύ περισσότερες δοκιμές ε, που θα πάρουν πολύ περισσότερο χρόνο, τότε μπορεί αυτό να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Ε, αυτό είναι το βασικό κριτήριο. Να μπουν στην αγορά, να βάλουν στην αγορά το νέο όχημα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί το κόστος κατασκευής ενός καινούριου μοντέλου είναι πολύ ψηλό και θέλουν γρήγορα να το αποσβέσουν. Ευχαριστώ πολύ. Για το μέλλον, πιστεύετε ότι με τον νέο κανονισμό θα έχουμε εγγύηση ότι θα έχει αίσιο μέλλον η αυτοκινητοβιομηχανία. Εγώ πιστεύω πως ε, υπάρχουν οι κίνδυνοι για την ε, βιομηχανία του ντίζελ. Γίνεται πολλή δουλειά για να περιοριστούν οι εκπομπές από τους ε, κινητήρες πετρελαίου και αν δούμε και το ποσοστό ανάπτυξης και μείωσης των εκπομπών είναι εντυπωσιακό το τι καταφέρνουν οι κατασκευαστές ακόμα και στις δοκιμές ε, υποπραγματικές συνθήκες περιορίζονται οι εκπομπές σε τεράστιο βαθμό. Τώρα βέβαια το ντίζελ έχει θέμα image. Δεν έχει καλή εικόνα και αυτό είναι πρόκληση γιατί υπάρχουν πολλές προκλήσεις ιδιαίτερα όσον αφορά την ποιότητα στο αέρα στα αστικά κέντρα για να δει κανεί γιατί έγινε τόσο δημοφιλές το ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό οδηγήθηκε, αυτό μάλλον ε, προκλήθηκε λόγω των ανησυχιών για το διοξείδιο του άνθρακα. Και υπάρχει άμεση συσχέτιση ανάμεσα στο πετρέλαιο και το διοξείδιο του άνθρακα. Ευχαριστώ κύριε Φιεμπράντη. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Κύριε Μπέρνς, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ερεύνα δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί οι αυτοκινητοβιομηχανίες ε, κλείνουν ε, την τεχνολογία αυτή στην πραγματική ζωή όταν είναι κατεστημένη, είναι μέσα στο κινητό. Γιατί να μην χρησιμοποιείται δηλαδή. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να ζητήσω από κάποιον που ήταν ε, μέσα στα πράγματα να μου το εξηγήσει. Και τι μου απάντησε. Μου είπε ότι τα βλέπετε λάθος τα πράγματα. Τα σκέφτεστε λάθος. Δεν τα σκέφτονται έτσι οι εταιρείε. Και μου είπαν λοιπόν ότι ο μοναδικός στόχος, ο πραγματικά μόνος στόχος των α, εταιριών κατασκευής αυτοκινήτων είναι να παράσουν ένα τεστ, ένα έλεγχο NEDC. Το τι γίνεται στην πραγματική ζωή μετά τον έλεγχο δεν έχει να κάνει τίποτα, δεν τους απασχολεί σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν απενεργοποιούν αυτή την τεχνολογία. Συμφωνείτε επί της αρχής με αυτή τη γενικότερη στοχοθέτηση των αυτοκινητοβιομηχανιών. Κοιτάξτε, δεν είμαι εγώ εταιρεία παραγωγής αυτοκινήτων, άρα δεν έχω άποψη. Πρέπει να περάσουν τις προδιαγραφές και τον έλεγχο. Και θα πρέπει να παράγουν τελικά αυτοκίνητα τα οποία να θέλει να τα αγοράσει και ο κόσμος. Άρα, σε τελική ανάλυση νομίζω ότι ναι, έχουν πολλά κίνητρα και πολλούς σκοπούς σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές, οι οποίες είναι περίπλοκες και πρέπει να τις ακολουθούν οι μηχανικοί τους. Αλλά ξέρουμε ότι η συμμόρφωση με τους είναι βασικό ζήτημα. Μία άλλη ερώτηση. Για κάτι που είπατε πιο πριν, σε ό,τι αφορά το συντελεστή συμμόρφωσης 2,1. Είπατε ότι αυτό ενδεχομένως να είναι δύσκολο να τον πετύχουν ως στόχο οι εταιρείες Κατασκευή αυτοκινήτων. Για εξηγήστε μα εννοείται για όλα τα αυτοκίνητα diesel, για τα πιο μικρά αυτοκίνητα diesel. Γιατί η τεχνολογία υπάρχει. Οι τιμέ ενδεχομένω να είναι λίγο πιο τσιμπημένες για τα μικρά αυτοκίνητα, αλλά θα μειωθούν δραματικά αν χρησιμοποιηθούν πιο μαζικά. Άρα πείτε μας, πού έγινε ακριβώς αυτή η πρόκληση. Το σχόλιο μου ήταν βασισμένο στις ε, τρέχουσες τιμές εκπομπών στο δρόμο σε σχέση με το 8 μιλιγκράμμα ανά χιλιόμετρο που, που προβλέπονται από τον νόμο και πάμπολες μελέτες καταδεικνύουν ότι είναι πενταπλάσιες, εξαπλάσιες οι εκπομπές, οι πραγματικές, στο δρόμο σήμερα. Άρα, το να περιορίσουμε το πενταπλάσιο σε 2,1 σημαίνει ότι ζητάμε από τους κατασκευαστές να μειώσουν τις εκπομπές τα 2 τρίτα. Είναι μεγάλη η εμπορική και η τεχνική πρόκληση σε ό,τι αφορά τα μεγάλα αυτοκίνητα, για παράδειγμα τα βαρέα οχήματα. Υπάρχουν κάποια ζητήματα, είναι πιο ακριβά. τα ελαφρύτερα αυτοκίνητα, τα οποία είναι μικρότερη αξία, έχουν άλλα ζητήματα να αντιμετωπίσουν σε ό,τι αφορά το κόστο των ε, αντίμετρων που θα πρέπει να λεφτούν. Είναι μεγάλη πρόκληση να περάσουμε από το εξαπλάσιο στο 2,1. Και τέλος, ο κύριος Eichhout. Ε, ναι, να συνεχίσω στο ίδιο πλαίσιο σε ό,τι αφορά τις τελευταίες ερωτήσεις και τη γενικότερη θεώρηση του θέματος. Μου έκανε εντύπωση το σχόλιο που κάνατε ότι οι εταιρείε παρασκευή, κατασκευής αυτοκινήτων θέλουν ακόμα να κατασκευάζουν καλά αυτοκίνητα. Από την άλλη, σας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι είναι πιο καλή η απόδοση του αυτοκινήτου όταν είναι ψυχρή η εκκίνηση από τη θερμή εκκίνηση. Γιατί το λογικό θα ήταν να είναι τα πράγματα καλύτερα με τη θερμή εκκίνηση. Αλλά αν το ξέρετε αυτό, και γι' αυτό δυσκολευόμαστε κι εμείς. Αν ξέρετε ότι τα 53 αυτοκίνητα τα οποία έλεγξε το Υπουργείο Μετακίνησης και Οχημάτων, 48 από τα 53 είχαν καλύτερα αποτελέσματα με την ψηφιακή κίνηση. 48 από τα 53. Πώς προκαλεί η έκπληξη, λοιπόν, το γεγονός ότι έχουμε αμφιβολίες για το ότι οι εταιρείε κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να κατασκευάσουν καλά αυτοκίνητα. Εσείς δηλαδή πώς έχετε πίστη και εμπιστοσύνη στο ότι κάνουν καλά τη δουλειά τους. Κοιτάξτε. Επειδή γνωρίζω και τα άτομα που συμμετέχουν στις εταιρείε αυτές, ξέρω τι ερωτήσεις μας κάνουν, ξέρω τι τους απασχολεί του απασχολεί να είναι νομιμή και κάνουμε πολλού ελέγχου, πολλά τεστ σε οχήματα που είναι ανάπτυξη ακόμα για να είμαστε βέβαιοι ότι θα περάσουν τα τεστ έγκριση τύπου όταν θα υποβληθούν προς έλεγχο. Ναι, αλλά όταν στην πράξη εκπέμπουν πενταπλάσιες, εξαπλάσιες ποσότητες α, αυτό είναι παράνομο δεν είναι παράνομο, γιατί το όριο ορίζεται σε έναν κύκλο ο οποίος είναι εντελώς παροχημένος. Αυτό ορίζει η νομοθεσία σε ό,τι αφορά το NDC. E ναι, αλλά αυτό αφορά μόνο την έγκριση τύπου και ο γενικότερα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον νόμο. Ο νόμος ορίζει κάποια όρια, ναι, αλλά τα όρια αυτά ορίζονται βάσει της ε, δοκιμής έγκρισης τύπου. Αυτό συζητάμε. Ότι η νομοθεσία δεν ανταποκρίνεται στι ανάγκε του πραγματικού κόσμου. Ναι, αλλά εδώ λοιπόν επανερχόμαστε σε θέματα κανονική χρήση. Γιατί αυτό λέει η νομοθεσία. Θα πρέπει να συμμορφώνεται σε κανονική, σε κανονική χρήση. Και αν είναι ασαφή η νομοθεσία, μα έχετε ρωτήσει ποτέ, έχετε ζητήσει ποτέ από κανένα στι Βρυξέλλε να σα διευκρινίσουν την νομοθεσία, γιατί είναι τόσο περίεργο αυτό που μα λέτε, που φαντάζομαι ότι θα έχετε ζητήσει διευκρινήσει, όπω είπα και προηγουμένως. Ε, γίνονται ε, συνεδριάσεις και υπάρχουν επιτροπές στα πλαίσια των συνδικαλιστικών οργανώσεων, γιατί είναι παροχημένος ο τρόπος μέτρησης στο πλαίσιο του NEDC για την έγκριση του τύπου. Είναι παροχημένος ο τρόπος διεξαγωγής των δοκιμών. Και πολύ απλά οι κανονισμοί αυτοί θα πρέπει να ενημερωθούν. Γίνεται βέβαια αυτό, αλλά αργά και βασανιστικά. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε άλμα από ένα αποτέλεσμα ελέγχου το οποίο δεν είναι κανονικό στο ότι όλοι είναι παράνομοι. Αυτά ορίζουν άλλωστε οι προδιαγραφές. Αν προδιαγράψουμε ένα κανόνα πολύ απλά, ο κόσμος προσαρμόζεται βάσει αυτό Ερώτηση, ναι, αλλά ξέρουμε ότι οι συσκευές αυτές οι διατάξεις αναστολή είναι παράνομες και ο μοναδικός τρόπος που μπορεί να πετύχουμε τα αποτελέσματα αυτά είναι το λογισμικό. Άρα αυτό τι είναι αν δεν είναι διάταξη αναστολής. Απλά έως τώρα δεν έχει κατανομαστεί αυτό ως διάταξη αναστολής. Εσείς πιστεύετε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, όπως είπα και προηγουμένο, προηγουμένως, αν υπάρχει κάποια τεχνική ανομαλία θα πρέπει να ερευνηθεί από τεχνική άποψη. Αυτό που δεν με βρίσκει σύμφωνο είναι το αυτόματο συμπέρασμα ότι πρόκειται για κάτι παράνομο. Μπορεί να υπάρχουν ελπεφανείς νόμιμες εξηγήσει, όπου οι κατασκευαστές ακολουθούν την νομοθεσία. Αν πρόκειται για κάτι ανεπιθύμητο, έμα θα πρέπει να διορθώσουμε τις προδιαγραφές και να πούμε ότι δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που επιθυμούμε πλέον οι προδιαγραφές και η νομοθεσία, άρα θα πρέπει να τροποποιηθούν, γιατί οι εταιρείε ε, θέλουν να είναι σύνομε. κανεί δεν θα θαυμάσετε τη Volkswagen για την καταστροφή που υπέστη. Ναι, ενδιαφέρουσα αυτή η άποψη, λέει η πρόεδρο, κυρία Μπέρνς. Ολοκληρώθηκε εδώ η ακρόασή μα και νομίζω ότι όλοι μα σα ευχαριστούμε για τι σαφεί σα απαντήσει. Μα βοήθησαν ιδιαίτερω. Και ως ε, συνήθως ε, θα υπάρχουν και κάποιες ερωτήσεις οι οποίες δεν απαντήθηκαν λόγω τεχνικών στοιχείων. Όσοι συνάδελφοι θέλουν να υποβάλουν άλλες γραπτές ερωτήσεις, μπορούν να το κάνουν αυτό μέχρι τις 17 Οκτωβρίου. Τα λέμε λοιπόν αύριο στις 9. Σας ευχαριστώ πολύ.